Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε στις 5 θα έρθει ο Επίτροπος για ανταλλαγή απόψεων και μέχρι τότε πρέπει να διεκπαιρεώσουμε τέσσερα σημεία της ημερήσιας διάταξης ε, και έχουμε ήδη κάποια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε πρόβλημα με την τσεχική διερμηνία. Μπορείτε να ακούτε. Μάλλον μπορείτε να μιλάτε, αλλά δεν μπορείτε να ακούτε τσεχικά. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Απαλλαγή 2013. Γενικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάρ' το Entwurf, δώσε στη... Moment. Oui, oui, Monsieur le Président, si vous permettez, je... Αν μου επιτρέπετε, μία διευκρίνηση, ένα διαδικαστικό. Πολλές φορές απουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις συνεδριάσεις μας. Σας έχω στείλει και σχετική επιστολή. Σας ευχαριστώ για την απάντηση και την αυρότητα. Αλλά καλό θα ήταν να επισημάνουμε αυτή την απουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσουμε να εμπλακεί πιο ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι στέλνει εκπροσώπους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάσεις. Δεν είμαι της ίδιας γνώμης. Εν πάση περιπτώσει, σημειώνω το σχόλιο σας, αν και έχω διαφορετική εντύπωση. Αν όντως ισχύει, είναι πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, σημείο 7, απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2013. Ε, αρμόδια κατ' Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Σύνταξη γνωμοδότησης ε, έχει δική μας Επιτροπή ε, με συντάκτη τον κύριο Γιάρ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και μάλιστα οι διάφορες επιτροπές οι αρμόδιες κατ' ουσίαν συμμετέχουν στην συζήτηση αυτή για τη χορήγηση απαλλαγής. Η έκθεσή μας στηρίζεται στην ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και στις ε, δικές μας έρευνες καθώς και τις συστάσεις του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, στον συντάκτη της γνωμάδας, τον κύριο Γιάρ, που έχει πείρα γιατί αναλαμβάνει εθίμοτυπικά κάθε φορά το θέμα της απαλλαγής. του δώσω το λόγο για να μας δώσει κάποια στοιχεία και να μας κατατοπίσει για την απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα παρουσιάσω την πρότασή μου ε, με μορφή γνωμοδότησης. Αρχίζω με τα πιο σημαντικά. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 9η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, παράκληση στους Κιώδης. 9 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, γιατί τίποτα δεν είναι τόσο καλό ώστε να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Δεύτερη παρατήρηση, ευθύ εξ αρχή. Πρώτη φορά γνωμοδοτεί η Επιτροπή μας για την απαλλαγή του προϋπολογισμού. Αυτό είναι καλό. Η υπεύθυνη Επιτροπή είναι η Επιτροπή Κοκομπού ε, δεν είχε ζητήσει παλιότερα γνωμοδότηση δική μας, τώρα το κάνουμε γιατί είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να γνωρίσουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που επηρεάζει άμεσα τους γεωργούς μας. Ακούγομαι, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Αρχίζω με έναν έπαινο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εντατικός διάλογος μεταξύ αν θέλετε του Κοκομπού, του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Κομισιόν από το 1999 και βέβαια ο γεωργικός τομέας είναι ε, από εκείνους που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά σφαλμάτων ε, σε άλλους τομείς. Ε, παλιότερα ήταν ακόμα χαμηλότερο το ποσοστό σφαλμάτων. Ίσως επειδή ε, δεν δεν, το ποσοστό δεν παρουσιαζόταν τόσο διεξοδικά. Ένα παρόμοιο σύστημα εντοπισμού και παρουσίασης ε, σφαλμάτων πρέπει να υπάρχει και αλλού στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην ε, Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, εγώ κατέγραψα 13 σημεία, σε 3 θα αποφανθώ, στο σημείο 4 όπου μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ποσοστών σφαλμάτων που παρουσίαζαν τα κράτη-μέλη και που ανακοίνωνε η Κομισιόν. Αν είναι σωστή η πληροφορία της Κομισιόν ε, και δεν είναι παράλογο, αν τα κράτη-μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά κάποια πράγματα, αυτό το ορίζουν δεν το ορίζουν ως φάλμα. Η Κομισιόν όμως αργότερα ε, παρουσιάζει άλλο ποσοστό σφάλματος. Ε, αν αυτό ισχύει θα δούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μειώνεται η διαφορά. Εγώ είμαι αισιόδοξο, έχω καλή πίστη, πιστεύω στο διάλογο μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών και θεωρώ ότι το ποσοστό σφαλμάτων θα ε, μειώνεται γιατί δεν θα γίνεται το ίδιο σφάλμα δύο φορές. Το επόμενο σημείο είναι το 11. Αυτό που μας ενοχλεί λίγο εμάς ε, είναι ότι η Κομισιόν και το, το ελεγκτικό συνέδριο ορίζουν διαφορετικά και παρουσιάζουν διαφορετικά τα σφάλματα. Το αιτιολογούν και οι δύο πλευρές, έχουν δηλαδή διαφορετικό σύστημα ε, παρουσίασης και αναφοράς, αυτό μπορεί να είναι αληθές και ο καθένας υπερασπίζεται το σύστημά του και λέει ότι δεν μπορούμε να αναμίξουμε τα δύο συστήματα. Εγώ όμως τονίζω στην έκθεσή μου ότι εμεί οι βουλευτές δυσκολευόμαστε ε, γιατί οι αισιόδοξοι παίρνουν τα κατώτερα ποσοστά, οι απεσιόδοξοι τα υψηλά. Καλό είναι όμως να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα. Να συμφωνήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι δύο ε, επί ενός ποσοστού σφάλματος. Ε, επίσης, θέλω μικρότερα προγράμματα που είναι στον πρώτο πυλώνα αυτή τη στιγμή να πάνε στο ποσοστό σφαλμάτων του δεύτερου πυλώνα. Γιατί? Διότι 80% των κονδυλίων είναι άμεσες ενισχύσεις, 20% στο δεύτερο πυλώνα. Τα μικρά προγράμματα ανεξάρτητα από τους λόγους, έχουν ποσοστό σφάλματος πάνω από το μέσον όρο. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε ε, ε, ότι ε, ο πρώτος πυλώνας για μας είναι πολύ σημαντικός για τη στρατηγική μας, γιατί βρίσκεται, είναι οι άμεσες ενισχύσεις και το ποσοστό σφάλματος θα πρέπει να ε, συνδεθεί με τον πρώτο πυλώνα και τις άμεσες ε, ενισχύσεις, γιατί εκεί έχουμε καλά αποτελέσματα. Ε, είναι ένα success story αυτό. Τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς, καλό είναι να τις παρουσιάζουμε χαμηλά ποσοστά ασφάλματος. Στο δεύτερο πυλώνα έχουμε ένα θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα για το γάλα στα σχολεία και τα φρούτα στα σχολεία επιτόπου, δηλαδή στον χρήστη, ε, δημιουργεί σφάλματα, οδηγεί σε σφάλματα. Και δεν φταίνε οι τελικοί καταναλωτές, αλλά η γραφειοκρατία. Αν μειωθεί η γραφειοκρατία, θα ε, είμαστε πιο ανθεκτικοί στα σφάλματα. Ε, αυτό αφορά και τα προγράμματα ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης. Ε, πολλές φορές η γραφειοκρατία εμποδίζει την υλοποίηση. Και Τέλος, θέλω λιγότερη γραφειοκρατική ευρωπαϊκή ε, γεωργική πολιτική. Και το απόγευμα που θα συζητήσουμε με τον Επίτροπο θα το πω αυτό. Γιατί η γραφειοκρατία επιβαρύνει ποικιλοτρόπως ε, και ε, μέσα από ε, τις, Βρυξέλλες επηρεάζει τα κράτη-μέλη, τους γεωργούς, την, ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη και επηρεάζει και τα ποσοστά σφάλματος. Ε, δηλαδή η γραφειοκρατία μόνο μειονεκτήματα συνεπάγεται. Ε, δεν... Δεν βρήκαμε ε, ένα παρασιτοκτόνο κατά της γραφειοκρατίας όπως τα διάφορα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μας. Εκεί έχουμε αποτύχει. Τώρα, το greening, το πρασίνισμα. Ε, εδώ έχω ανάμεικτα συναισθήματα, είναι καινούριο σύστημα. Δεν είναι απαλλαγμένο από γραφειοκρατία και νομίζω ότι με την εισαγωγή του greening θα αυξηθούν και τα ποσοστά σφάλματος στα κράτη-μέλη. Και αυτό μας δημιουργεί δυσκολίες ερμηνείας, γιατί οι κοινοί γνώμοι λένε τι κάνουν ε, ε, μοιράζουν χρήματα στους γεωργούς αλλά τα ποσοστά ασφάλματος ε, αυξάνονται. Το greening λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το εισαγάγουν και να το εφαρμόσουν με τρόπο που να μην επιδέχεται σφάλματα. συνολικά βέβαια συστήνω απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Ωραία για συζήτηση. Ο κύριος ε, Ρόντε ζήτησε πρώτος το λόγο σε αυτό το γύρο. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάρ για την ενεργασία του αυτή επί του προπολογισμού. Καταρχήν, στην ομάδα των φιλελευθέρων είμαστε υπέρ του σχεδίου αυτού. Δύο ερωτήσεις. Προτείνεται ε, τη χρηματοδότηση σχολικών προγραμμάτων να χρηματοδοτούνται στο δεύτερο και όχι στον πρώτο πυλώνα. Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το γιατί και ρωτώ. Δεν υπάρχει ένας κίνδυνος τα ε, κονδύλια της αγροτικής πολιτικής να πηγαίνουν για άλλους σκοπούς στα κράτη-μέλη, να χρησιμοποιούνται αλλού. Και για τον έλεγχο των σφαλμάτων, για το στόχο βέβαια δεν διαφωνεί κανείς εδώ στην Επιτροπή, αλλά πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί το πρόγραμμα στην πράξη. Ε, δηλαδή στους οργανισμούς πληρωμών να πάνε σε κεντρικό επίπεδο υπάλληλοι της Κομισιόν ε, κατά τα άλλα συμφωνώ με την προσέγγισή σας, αλλά πάνω σε αυτό θα ήθελα κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Πέτερ για τη δουλειά του. Υπάρχει ύψιστη σύγκληση και συμφωνία με αυτά που είπε. Το θέμα της απλούστευσης είναι κεντρικό ζήτημα και είναι και το νέο διακύβημα της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Θέλουμε να είναι πιο απλή η διαδικασία και αντί περιπλέκεται. Για το σημείο 7 υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δυνατότητα ε, της ε, μετάθεσης των προγραμμάτων της εμβελίας στο δεύτερο πυλώνα. Υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει το αντικείμενο και επειδή κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι πάνε πλέον από εθνική διαχείριση σε περιφερειακή διαχείριση, που είναι για τη χώρα μου. Και αυτό θα μπορούσε να προξενήσει ε, δεκάδες διαφορετικά προγράμματα και αντί να πλουστεύσουμε περιπλέκουμε τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το πρασίνισμα, συμφωνώ με σένα, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και ελπίζω να μπορέσουμε να τα πλουστεύσουμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Α, συγγνώμη, ο κύριος Μπούντα έχει απομείνει στον κατάλογο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Γιάρ. Και είμαι βέβαιος ότι θα σχολιάσουμε αυτό το θέμα και αργότερα στη συζήτηση που θα έχουμε με τον ε, Επίτροπο, γιατί χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, ε, τουλάχιστον στον greening, στο πρασίνισμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ε, στις εκτιμήσεις της Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν να διαλευκάνουμε τις αιτίες αυτών των διαφορών και να διευκρινίσουμε τη σχετική νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 9, ζητά από τους εξεματούχους ε, της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν τον έλεγχο στη θέση των αξιωματούχων κρατών μελών. Νομίζω ότι μια τέτοια ανάθεση αρμοδιοτήτων θα ενισχύσει τη δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και όχι να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Δεν ζητά άλλος κανείς το λόγο, οπότε θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Μάγκελε, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να επενέσω την Επιτροπή, διότι για πρώτη φορά καταπιάστηκε με το δύσκολο αυτό θέμα της απαλλαγής και το ποσοστό σφαλμάτων στην κοινή αγροτική πολιτική. Εμείς στις υπηρεσίες της Κομισιόν πάντοτε αντιμετωπίζουμε το δίλημα από τη μια πλευρά να εξυπηρετήσουμε την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, την Κοκομπίου και να δώσουμε πληροφορίες και πολλές φορές δεχόμαστε από αυτούς επικρίσεις και εσείς πολλές φορές βέβαια μας επικρίνετε, αλλά εσείς λέτε πράγματα κατά της ε, γραφειοκρατίας των αυστηρών ελέγχων που κάνουν να υποφέρουν οι γεωργοί. Αυτή τη θέση λοιπόν που εκφράζεται, καλό είναι που περνάει στην έκθεση και παίζει ρόλο στην απαλλαγή. Η έκθεση νομίζω ότι έχει πολλές πολύτιμες πληροφορίες και εκφράζει τις θέσεις της Επιτροπής πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες τεχνικής φύσης διορθώσεις που θα πρότεινα να γίνουν. Μπορώ να το κάνω άμεσα με τον εισηγητή. Α, το έχω κάνει ήδη. Υπάρχουν κάποια νούμερα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις τώρα για σημεία που ετέθησαν και εδώ στη συζήτηση. Καταρχήν το σημείο 4 που ανέφερε ο κύριος Γιάρ, ο δόκτωρ Γιάρ, δηλαδή η λάθος αναφορά από τα κράτη-μέλη. Εμείς στην Κομισιόν δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι εκ προθέσεως δίνουν λάθος νούμερα τα κράτη-μέλη και το ελεγκτικό συνέδριο λέει τα ίδια. Διαπιστώνουμε όμως ότι οι έλεγχοι που γίνονται στα κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετά σωστοί για να εντοπίσουν όλα τα προβλήματα. Και όταν πάει επί τόπου το ελεγκτικό συνέδριο ή εμείς με τους ελέγχους βλέπουμε πρόσθετα σφάλματα και δυσκολίες και στις εθνικές ε, στατιστικές και στα ποσοστά σφάλματος στα εθνικά δεν περιλαμβάνονται. Δεν είναι λάθος ο τρόπος αναφοράς, αλλά η βασική δουλειά που γίνεται επί τόπου δεν είναι καλή και προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο θέμα είναι το υπαριθμόν 6 της έκθεσης, όχι το 7, που αναφέρεται ότι μια λύση θα ήταν ίσως τα μικρότερα προγράμματα, αναφέρθηκε το γάλα στα σχολεία, να πάνε από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Ε, Δόκτωρ Γιάρ, κατάλαβα ότι δεν θέλετε μετατόπιση της πολιτικής στο δεύτερο πυλώνα, μόνο τη μετατόπιση στο δεύτερο πυλώνα των ε, μέτρων για τον υπολογισμό των σφαλμάτων. Αυτό βέβαια είναι ε, από πολιτικής άποψης τελείως διαφορετικό από το να περάσει η πολιτική. Αν πρόκειται για τη μετατόπιση των ποσοστών σφάλματος θα έχουμε μεγάλα προβλήματα γιατί το ποσοστό σφάλματος ως Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου ε, καταρτίζεται για συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και για τον δεύτερο πυλώνο προϋπολογισμός είναι ένα ειδικό κομμάτι του προπολογισμού που έχει το δικό της ποσοστό σφάλματος και το πρώτο πυλώνας ε, επίσης είναι ένα κομμάτι και το ελεγκτικό συνέδριο ε, υπολογίζει ένα ποσοστό σφάλματος εκεί για τα, τις άμεσες ε, ενισχύσεις και τα μέτρα για την αγορά. Από τεχνική άποψη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών μου φαίνεται ότι δεν θα το δεχτούν. Το επόμενο είναι το 9, δηλαδή να είναι επικεφαλής υπάλληλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνη για τους οργανισμούς πληρωμών όταν γίνονται σφάλματα διαχείρισης. Ε, και προσωπικά και οι Κομισιόν θεωρούμε ότι δημιουργούνται έτσι νομικά προβλήματα γιατί πώς είναι δυνατόν να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη κοινοτικούς ενωσιακούς υπαλλήλους δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο, θα έπρεπε πρώτα να δημιουργηθεί. Και αν θα είχε ευκαιρία κάτι τέτοιο να περάσει από το Συμβούλιο, δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, αλλά αμφιβάλλω. Το δεύτερο θέμα όμως ε, ε, αφορά και τους φορείς. Το 5% των θέσεων στην Κομισιόν θα καταργηθούν άμεσα. Ε, αν στείλουμε έναν υπάλληλο θα έπρεπε να βρούμε 82 θέσεις ακόμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ούτε ένας θα ήταν αρκετός κατά πάσα πιθανότητα. Θα έπρεπε να πάνε και άλλοι. Σκεφτείτε το. Με τη, στη σημερινή συγκυρία γίνεται κάτι τέτοιο. Και τρίτο και σημαντικότερο. Η γεωργική διοίκηση και διαχείριση λειτουργεί με βάση την επιμερισμένη διοίκηση. Δηλαδή η ευθύνη για τη διεξαγωγή της αγροτικής πολιτικής επιμερίζεται μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών, όπου η Κομισιόν μέσω του προπολογισμού διαθέτει τα κονδύλια, υποβάλλει τις διατάξεις ε, που θα ε, εγκριθούν από τον νομοθέτη και κάνει μετά πράξεις και εκτελεστικές και κάνουν μετά την διαχείριση τα κράτη-μέλη. Αν πάνε στους οργανισμούς πληρωμών υπάλληλοι της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαλύεται η επιμερισμένη διαχείριση και η Κομισιόν θα είναι νομικά υπεύθυνη για κάτι το οποίο όμως δεν το διαχειρίζεται εκείνη επιτόπου. Και αναγκαστικά θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να μην είναι υπεύθυνα. Και ποιος θα είναι υπεύθυνο και αν οι έλεγχοι δεν λειτουργούν. Ε, θα ήταν αδιέξοδο κάτι τέτοιο και απευθύνω έκκληση να το ξανασκεφτείτε. Ε, τώρα, ε, το 11, δύο έχω ακόμα να αναφέρω, για τα διαφορετικά ποσοστά σφαλμάτων. Πράγματι, έχουμε διαφορετικά ποσοστά και εφαρμόζουμε διαφορετικές μεθόδους. Το ελεκτικό συνέδριο έχει ένα ποσοστό σφάλματος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ένωσης για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Ε, ξέρετε πόσο, ξέρουμε δηλαδή πόσο είναι το ποσοστό σφάλματος για τα μέτρα αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις αφενός και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης από η Κομισιόν πάει να υπολογίσει μέχρι το επίπεδο του κάθε οργανισμού πληρωμών, ε, χωριστά ε, στα τρία αγροτική ανάπτυξη, άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγοράς για να ξέρουμε έτσι που είναι τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Στόχος μας δεν είναι πρωτίστως δηλαδή να βοηθήσουμε το κοινοβούλιο για να απαλλάξει την Κομισιόν. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Θέλουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που διαπιστώνουμε επί τόπου να τα καταπιαστούμε με τρόπο αποτελεσματικό μαζί με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μέθοδος διαχείρισης. Αν πάμε στο στατιστική μέθοδο του ελεγκτικού συνεδρίου και αν αυτό θέλαμε να το κάνουμε σε επίπεδο οργανισμού πληρωμών θα έπρεπε να έχουμε ακόμα 2.000 ε, με 3.000 περισσότερους ελεγκτές αδύνατον. Ε, έχουμε διαφορετικά σημεία εκκινήσεως. Και γι' αυτό τα συστήματά μας μπορούν να συνυπάρχουν. Γιατί δεν οδηγούν αναγκαστικά σε πολύ διαφορετικά αποτέλεσμα. Το 2013 για τις άμεσες πληρωμές είχαμε σε επίπεδο κομισιών ποσοστό σφάλματος 2,32% και το ελεγκτικό συνέδριο ήταν 2,4% ε, σε νοσιακό επίπεδο. Κοντά είμαστε. Πρόκειται δηλαδή για διαφορές που αφορούν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το, το greening τώρα, το πρασίνισμα, αυτό είναι νέο μέτρο προφανώς. Κάθε νέο μέτρο οδηγεί νομοτελειακά σε κάποιους φόβους, σε κάποιες αβεβαιότητες. Από την άλλη πλευρά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικότερα για να ε, προχωρήσει σωστά με τη μεταρρύθμιση των άμεσων ενισχύσεων έχει φτιάξει ειδικό τμήμα με 18 υπαλλήλους που ε, σκοπό έχουν από κοινού με τα κράτη-μέλη να επεξεργαστούν τους εφαρμοστικούς κανόνες, να κάνουν διαβουλεύσεις και αν υπάρχουν αμφιβολίες να απαντούν και να δίνουν ερμηνεία. Το feedback ε, είναι πολύ καλό από τα κράτη-μέλη, πολύ θετικό και νομίζω ότι μέχρι την αρχή, τα μέσα της επόμενης χρονιάς, εν λήξη προθεσμία αιτήσεων μέσα Μαΐου, ε, θα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σαφήνεια σχετικά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τα κράτη-μέλη ε, έχουν επενδύσει στις μεταρρυθμίσεις αυτές εκατομμύρια ευρώ. Ένα κράτος μέλος είπε ότι στήχησε 20 εκατομμύρια ευρώ ε, το νέο σύστημα. Αυτά δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουν, να εξελιχθούν. Και πρέπει επίσης να σημειώσω ότι με την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίστηκε να μην, να υπάρχουν κυρώσεις τα πρώτα δύο χρόνια του, στο πρόγραμμα Greening, αλλά να αρχίζουν με, οι κυρώσεις τον τρίτο χρόνο όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες, οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής μας, ο Πίτερ Γιάρ. Ο κύριος Γιάρ. Ε, ευχαριστώ. Συνοψίζω τις παρεμβάσεις και προτείνω τροποποίηση σε τρία σημεία ε, και θα τα επεξεργαστούμε από κοινού μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Πρώτο σημείο, το σημείο 7. Εδώ πρόκειται για την μετατόπιση του ποσοστού σφάλματος. Αυτό τεχνικά δεν γίνεται. Να συμφωνήσουμε λοιπόν, να απευθύνουμε σαφή έκκληση στην Κομισιόν, ώστε τα προγράμματα, τα λεγόμενα μικρά προγράμματα, να τα απαλλάξει από τη γραφειοκρατία, γιατί το πρόγραμμα ε, για τα σχολεία ε, στηρίζεται σε καλές προθέσεις, αλλά έχει τόσο γραφειοκρατία που δεν εφαρμόζεται τουλάχιστον στη Γερμανία σε όλες περιφέρειες. Για το γάλα στα σχολεία είναι πιο οικονομικό να αγοράζει κανείς το γάλα από το σούπερ μάρκετ για τα σχολεία παρά να λειτουργεί το πρόγραμμα. Άρα κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να καθίσουμε να δούμε τι είναι, να μειωθεί η γραφειοκρατία και θα μειωθούν και τα ποσοστά ασφάλματος και θα εφαρμόζονται και περισσότερο. Οπότε μέχρι 9 Δεκεμβρίου καλό είναι εδώ να βρεθεί μια διατύπωση. στο σημείο 9, σωστό. Και εγώ προτείνω ε, τροποποίηση. Πρόκειται για το εξή. Αν ένα οργανισμό πληρωμών ε, επικριθεί επανειλημμένα από την Κομισιόν ότι ο οργανισμός, ο οργανισμός δεν παρουσιάζει ποσοστό σφάλματος, ενώ η Κομισιόν όταν πάει ε, βρίσκει πολλά λάθη και αν αυτό ε, συμβεί επανειλημμένα, τότε θα έπρεπε να ε, μπορεί κανείς να αποσύρει την πιστοποίηση από τον οργανισμό πληρωμών. Αν την κλείσει τέλος πάντων δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Και θα πρέπει να βρεθεί μια διατύπωση, ούτως ώστε αν, όταν δεν ανάψει κόκκινο, όταν ανάψει πορτοκαλί ή κίτρινο φως, να ε, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα. Δηλαδή δεν θα είναι ε, υποκατάσταση, δεν θα έρχεται δηλαδή ε, ως αντικαταστάτης ε, ή ως φορέας λήψης αναγκαστικών μέτρων ή κομισιών. Πάντως θα πρέπει να γίνει κάτι για τους οργανισμούς αυτούς. Θα το αναδιατυπώσω. Τώρα το 11, μια καλύτερη διατύπωση σχετικά με τα διαφορετικά ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται γιατί είναι η μέθοδος διαφορετική. Καλό θα ήταν να προσεγγίσει το ένα το άλλο. Θα κάνω καλύτερη διατύπωση. Δεν είναι ωραίο τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν διαφορετικά ποσοστά. Ε, ε, ε, δεν είναι εύληπτο το σύστημα έτσι. Ε, θα είμαι ευγνώμων για τις προτάσεις που θα μου υποβάλλετε. Με τους συναδέλφους θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση του 7 και του 11 ίσως. Ε, θέλω όμως και άλλες προτάσεις, δηλαδή πολύ θα χαρώ να έχετε ιδέες και να μου τις υποβάλλετε μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις 9 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Ωραία. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Είδαμε και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και τις προθεσμίες. Οπότε διεκπαιρεώσαμε το σημείο 7 και περνάμε στο 8. Ε, ζωοτεχνολογικές και γενεαλογικές συνθήκες για εμπόριο και εισαγωγές στην Ένωση ζώων, ε, ζώων αναπαραγωγής και γενετικού υλικού και προϊόντα και ένα υλικό. Έχουμε δύο νομοθετικές προτάσεις. Ο στόχος της ζωοτεχνικής ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διευκόλυση του εδοκινοτικού ελεύθερου εμπορίου και η διευκόλυνση των εισαγωγών ζώων αναπαραγωγής και του γενετικού τους αναπαραγωγικού υλικού. Και επίσης ε, η ε, διατήρηση προγραμμάτων αναπαραγωγής και προγραμμάτων διαφύλαξης των γενετικών πόρων προκειμένου να διατηρηθούν όλες οι φυλές που υπάρχουν στην Ευρώπη οι κράτους των ζώων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα η δεύτερη πρόταση αφορά κάποιες τεχνικές τροπολογίες. Ουσιαστικά θέλουμε να διαγράψουμε τον όρο ζωοτεχνικός σε τρεις ε, από τις υπάρχουσες οδηγίες. Το θέμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ε, για το νέο κανονισμό που αφορά τους επίσημους ελέγχους. Και για τις ε, δύο περιπτώσεις η συγκητής μας είναι ο Μισελ Νταντά. Θα εξετάσουμε από κοινού τα δύο θέματα. Κύριε Νταντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως είναι αλληλένδετες οι δύο εκθέσεις γιατί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συγκεράσει σε ένα κείμενο διατάξεις που υπήρχαν σε διάφορα νομοθετικά κείμενα ανά ε, και αφορούν το θέμα του το και γενετικό υλικό. Θέλουμε έτσι να διευκολύνουμε το ενδοκινοτικό εμπόριο και κυρίως ε, να καταστήσουμε πιο αξιόπιστα τα στοιχεία για την, για την γενετική βελτίωση των ζώων αναπαραγωγής. Κάποια τεχνικά σημεία ε, θα τα σχολιάσω και θα καταθέσω και προτάσεις και επίσης ε, να σας πω ότι κάποιοι ορισμοί που υπάρχουν στο κείμενο θα πρέπει να διευκρινιστούν για να ξέρουμε ότι μιλάμε όλοι για το ίδιο πράγμα και να υπάρχει συνεννόηση ως προς αυτό. Υπάρχει ένα ιδιάζον θέμα για τα υποειδή, για τις φυλές υποειδών. Εκεί δίστανται οι απόψεις, γιατί η επιλογή των ύπων γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα γενεαλογικά βιβλία που έχουμε την Ευρώπη κρατώνται από διεθνείς οργανισμούς που έχουν διοικητικό συμβούλιο και στο οποίο συμμετέχουν, εκπροσωπούνται όλες οι χώρες στις οποίες υπάρχει αυτή η ράτσα, αυτή η φυλή λοιπόν. Πρόκειται για ιδιάζουσα κατάσταση για τα υποειδή λοιπόν. Το κείμενο αυτό συζητήθηκε στον τριμερή διάλογο με συμμετοχή του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και αφορά τους επισήμους ελέγχους ε, περιμένουμε έκβαση την επόμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου θα συμπεριληφθούν μαζί με τις προτάσεις μας στην πρόταση κανονισμού που εξετάζουμε. Θα ήθελα να επιμείνω σε ένα κυρίω θέμα, το θέμα της αξιοπιστίας των δεδομένων. Γιατί σε ό,τι αφορά τη γενετική βελτίωση, τα ζώα αναπαραγωγής περιλαμβάνονται σε βιβλία και μητρό. Όταν θέλουμε να ξέρουμε πώς ε, ε, καταρτίζονται αυτοί οι δείκτες ε, σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση αυτών των δικτών στις διάφορες χώρες. ώστε ένας σταύρος αναπαραγωγής στη Γερμανία, για παράδειγμα, να θεωρείται το ίδιο και στην Αυστρία, παρόλο που μπορεί το γενετικό επίπεδο, το μέσο γενετικό επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Επίσης, ένα ζώο αναπαραγωγής ε, θα πρέπει να ξέρουμε πότε υποβαθμίζεται στην ΑΒ χώρα. Και έχουμε και τους αγοραστές εκτός της Ένωσης, γιατί δεν μιλούμε εδώ μόνο για δοκιματικές συναλλαγές. Εμείς προ... προμηθεύουμε ολόκληρο τον κόσμο με γενετικό υλικό, με υλικό αναπαραγωγής. Οπότε οι αγοραστές μας, οι πελάτες μας θα πρέπει να είναι σίγουροι για την αξιοπιστία των ε, ζώων αναπαραγωγής που αγοράζουν. Επίσης, ε, προτείνεται μια σειρά και καταξιοδότηση πράξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι παραδοσιακά καχύποπτο απέναντι στις καταξιοδότησεις πράξεις και η έξοδος τους από την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ μας κατέστησε ακόμη πιο δύσπιστους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού της κατεξουδότηση πράξη, Παρόλο που θεωρούμε ότι με κάποιες από αυτές θα πρέπει να αφήσουμε κάποια διακριτική ευχέρεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευρύνει τον κανονισμό και να περιλάβει κάποια άλλα είδη που δεν είναι ε, τα βασικά είδη στην Ευρώπη. Κάποια είδη πουλερικών, για παράδειγμα, κάποιες φυλές που να το πολύ περιορισμένα, μικρές φυλές στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάντως και τους και ηγητές για τη συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχίσουμε να έχουμε. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες θα συναντήσω και τους δύο-τρεις και ηγητές που δεν ε, συνάντησα ακόμη. Το κείμενο είναι αρκετά περίπλοκο γιατί έχει ιδιαίτερα τεχνικές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάντως για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Άρχεται η συζήτηση. Ο κύριος Φεράν ζήτησε το λόγο πρώτα. Παρακαλώ κύριε Φεράν. Φεράν. Φεράν. Uh, ευχαριστώ πολύ. Όχι εγώ. <laughs> Euh, λοιπόν, προτείνεται ένας νέος κανονισμός που αφορά τα ζωοτεχνικά θέματα και αντικαθιστά πολυάριθμους ισχύοντες κανονισμούς. Θα είμαι λακωνικός. Νομίζω ότι το να εξευρωπαίσουμε όλα αυτά τα ζώα θα θέσει σε κίνδυνο την κληρονομιά των ζώων που επένδυσαν πολλά χώρες όπως η Γαλλία για να διατηρήσουν τις ε, διάφορες ράτσες των ζώων και την ποικιλομορφία. Θα είναι πολύ δαπανηρός ο κανονισμός και η εφαρμογή του όσον αφορά τις ε, ράτσες που έχουν πολύ μικρό αριθμό ζώων και που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και ο των εγκεκριμένων οργανισμών για την έγκριση των διαφόρων ζώων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση της κληρονομιάς, της ζωικής. Είναι ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση του ζωικού κεφαλαίου προς όφελος μιας δράκας πολυεθνικών που αφορά την επιχείρηση του τομέα της αγροβιτικής βιομηχανίας. Εάν τροποποιήσουμε ή καταργήσουμε τον ε, ισχύοντα κανονισμό, όπως αναφέρεται στο σημείο 8, νομίζω ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Ντάντα για τα όσα μας είπε, για τις εξηγήσεις που μας έδωσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για, τους δύο, για τα δύο χαρτοφυλάκια τα οποία είναι αλληλένδετα εκτιμώ πολύ τα όσα έκανε. Ο κανονισμός προσπαθεί να ομαδοποιήσει διάφορους ε, τομείς νομοθεσίας δεσμευτικής για τα κράτη-μέλη κυρίως τους επισήμους ελέγχους στον ζωτεχνικό τομέα που έλεγχος αυτός θα είναι στα χέρια των αρμοδίων υπηρεσιών των αρχών που είναι υπεύθυνε για αυτά τα θέματα σε κάθε κράτος μέλος. Το σχέδιο κειμένου σέβεται τις αρχές της ενώσεως αλλά κατά κάποια έννοια θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα κυρίως όσον αφορά την υστέρηση που υπάρχει μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Εκτινοτρόφοι και διάφορες οργανώσεις ε, των κτηνοτρόφων βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και επίπεδα πλούτου θα έλεγα στα νέα κράτη-μέλη τα προγράμματα έχουν μείνει κάπως πίσω και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Με τη βοήθεια του κυρίου Νταντά είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Μιλάμε για δύο προγράμματα, συζητούμε τις δύο σχετικές εκθέσεις. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις επιθυμίες των κτηνοτρόφων. Αυτές οι τέσσερις οδηγίες να συμπυκνωθούν σε ένα νομοθέτημα. Αυτό το νομοθέτημα θα είναι πιο εύληπτο και θα είναι πιο εύκολο να συμμορφωθούν με αυτό. Χαιρετίζω λοιπόν τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι αξιέπαινη η προσέγγιση της και θέλω να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερα τον κύριο Ταντέν για τις εξηγήσει που μου έδωσε σε μια προηγούμενη συνάντηση και προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία μαζί του. Dziękuję. Proszę posła Federli. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Νταντέν. Σας ευχαριστώ κύριο Νταντέν για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Αυτό που επεξεργαζόμαστε, προχωρημένο το θέμα και έχω κάποια θέματα να θίξω. Διατείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές, συγχωνεύοντας τα τέσσερα κείμενα. Να έχουμε υπόψη όμως ότι κάποιοι, για κάποιους οργανισμούς κτηνοτρόφων και αναπαραγωγή ζώων ίσως να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ε, υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τους επισήμους ελέγχους που θα διενεργούνται. Αυτό είναι θετικότατο. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το νομικό πλαίσιο της επισήμου ελέγχους που έχουμε πάρει από την νομοθεσία που είχε κατασκευαστεί, που είχε θεσπιστεί για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπικάλυψη και δεν πρέπει να δεσμεύουμε υποβολικά τους ε, γεωργού και του κοινοτρόφου. Πλευρά Άλντα ανησυχούμε για τι τις στην πράξη, τον αριθμό αυτών. Ε, πολλά θα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, χωρί να έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Άρα χρειάζονται και άλλες συζητήσεις από αυτού, να δούμε πως υπάρχει άλλη λύση. Ίσως υπάρχει πρόβλημα της ορισμούς. Το αναπαράγω ή μεγαλώνω ζώο σημαίνει, η λέξη breed η αγγλική σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διάφορες χώρες. Και πρέπει να ακούσουμε και τους αρμόδιους οργανισμούς ε, να αποφύγουμε να τους δημιουργήσουμε προβλήματα. Θέλουμε τα τέσσερα διαφορετικά πλαίσια να τα κάνουμε ένα και να γίνουν πιο συνεκτικοί οι κανονισμοί και πιο εύληπτοι για τους κτηνοτρόφους. Αυτά έχω να πω σαν πρώτες παρατηρήσεις από πλευράς της ε, πολιτικής ομάδας της ΑΛΤΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλές οργανώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων προβληματίζονται από αυτό. Έχουν μιλήσει μαζί μου, με εξέφρασαν και κάποιες απορίες που θα σας διαβιβάσω. Πρώτα απ' όλα, η δομή των διαφόρων φορέων που αναφέρονται, που εφαρμόζουν τα προγράμματα αναπαραγωγής, η δομή τους άλλαξε. Συγγνώμη κυρία μου, κάτι... Είχαμε ένα πρόβλημα με την γαλλική διερμηνία και επειδή ο εισηγητής μας είναι Γάλλος ε, πρέπει να ακούσει τα σχόλιά σας. Μπορείτε τώρα να συνεχίσετε. Καλώς. Συνεχίζω. Εντάξει, ακούγονται τα γαλλικά. Ωραία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να, του να θέσω αυτά τα θέματα. Έχει αλλάξει ε, πολύ ε, ο κανονισμός, έχουν αλλάξει οι δομές για τα προγράμματα τα αναπορογικά σε κάποιες χώρες. Σε κάποιες χώρες έχουν εφαρμοστεί τα αναγκαία μέτρα, αλλού όχι. Υπάρχει ίσως ενδεχόμενο να εφαρμόσουμε με ευελιξία τα μέτρα. Και τι γίνεται με την αναπαραγωγή των χείρων και την αναγνώριση της σχετικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί για την αναπαραγωγή των χείρων και την ανατροφή των χείρων και για τα βοηδή να είναι εντελώς διαφορετικοί. Τι συγκρίσεις υπάρχουν μεταξύ αυτών. Και τι γίνεται με την καθαρότητα, την γενετική των διαφόρων ζώων. Γιατί πολύ συχνά δεν είναι πολύ εύκολο να εντοπίσει κανείς τα καθαρά γονίδια και θα πρέπει να εξετάσουμε τους ε, ορισμούς αν θέλουμε να θεσπίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Ξέρω ότι είναι τεχνική φύση αυτό, αλλά θα πρέπει να τα εξετάσουμε για να έχουμε μια νομοθεσία η οποία να μπορεί να λειτουργήσει τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Νταντά, για τα σχόλιά του και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση κανονισμού. Είναι σίγουρα σημαντικό και απαραίτητο να διευθετήσουμε το θέμα αυτό και είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Μιλούμε για τη γενετική πρόοδο, για την εκτροφή των ζώων, για την αναπαραγωγή. Και για να έχουμε γενετική πρόοδο θα πρέπει να γίνει σωστή, αυστηρή επιλογή του αναπαραγωγικού υλικού και προσοχή στη διαδικασία αναπαραγωγής και στην εκτροφή. Υπάρχουν ε, πολλές δυσκολίες ε, κατά την εφαρμογή του κανονισμού αυτό από τα κράτη-μέλη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία εναρμόνιση των μητρών ε, των διαφόρων φυλών. Ιδιαίτερα για τα καθαρό αίμα ζώα, γιατί θα πρέπει η εκτροφής να είναι σίγουρη για την ποιότητα και το γενεαλογικό και γενετικό υλικό των ζώων τους. Θέλουμε την δέουσα προστασία για τις φυλές που έχουμε τώρα και για αυτές που θα δημιουργηθούν και στο μέλλον με υβριδικό τρόπο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΜΚΟ, τον κύριο Βόλγαταν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Η πρόταση είναι αρκετά σαφής κατά την άποψή μας. Είναι αναδιατύπωση υφιστάμενης νομοθεσίας που ισχύει εδώ και 30 χρόνια. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη το σύνθημα καλύτερη νομοθεσία, απλούστευση. Βασιστήκαμε και στην εμπειρία μας των, τις τελευταίες 30 και διαφόρων θα πρέπει λοιπόν οι εταιρείε της αναπαραγωγής των ζώων να λειτουργούν σωστά στην ιστορική αγορά. Θέλαμε λοιπόν η ενιαία αγορά για την αναπαραγωγή των ζώων και για τη διατήρηση των διαφόρων ζώων και για, τα υβριδικά, για τους υβριδικούς χείρους όπως αναφέρθηκε να λειτουργεί σωστά. Ένα καθαρό ζώο σε μια χώρα θα αναγνωρίζεται σαν καθαρό ζω και σε άλλο κράτος μέλος. Όπως το σαρολέ, το σαρολέ στη Γαλλία πρέπει να θεωρείται σαρολέ και στο Βέλγιο και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν εκείνοι που διατηρούν και ανατρέφουν τα, διατρέφουν τα α, καθαρό αίμα να αναγνωρίζονται και να πληρούν υψηλά κριτήρια ώστε να έχουμε υψηλά επίπεδα εκτροφής των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έπρεπε το δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσίας για εκείνες τις εταιρείε εκτροφής να ε, καθιερώνονται και να αναγνωρίζονται από τα κράτη-μέλη. Κάποιοι ανέφεραν και τους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν διενεργούνται απευθείας στα ζώα, αλλά στην εταιρεία που έχει τους τάβλους, στην επιχείρηση και καθορίζουν εκείνη τα καθαρό αίμα. Τι είναι καθαρό μοζό. ζώο. Δεν θέλουμε εμείς να καθορίσουμε εδώ ή στα κράτη-μέλη στη δίκη των κρατών μελών. Τι είναι ένα καθαρό αίμα ζώο. Η στα κρατη μελη στη δικη των κρατων μελων τι ειναι ενα καθαρο αιμο ζωο η εταιρεία θα πρέπει να το ορίζει και να πληρεί κάποιους όρους για να λειτουργεί σωστά. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τα σπάνια είδη και τη γενετική ποικιλομορφία του ζωικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κύριε Πρόεδρε, με αυτά θα πω ότι με τα χαρά σας συνεργαστούμε με τον εισηγητή, θα είμαστε στενή ε, συνεργασία μαζί του για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε συγκεκριμένη υπόθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος και πάλι στον εισηγητή μας, τον κύριο Νταντά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και να πω ότι ε, μεριμνούμε όχι για να περιπλέξουμε τα πράγματα αλλά για να τα διευκρινίσουμε. Όπως αναφέρθηκε εδώ και 30 χρόνια είχαμε διάφορα κείμενα, πολλές ε, νομοθετικές διαστάσεις, ε, διαφορετικές είδος. Φυσικά δεν θα παραβλέψουμε τη διαφορετική οργάνωση σε κάθε χώρα αλλά δεν θα πρέπει να είναι επιζήμια αυτή η διαφορά. Γι' αυτό και οι οργανώσεις και εκτροφής ε, θα πρέπει να έχουν στόχο την προσφορά αξιόπιστων δεδομένων. Θέλουμε διαφανή, ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα. Αυτό είναι κοινό μέλημα για όλους. Έχουμε φυσικά γενετικό δυναμικό για διάφορες φυλές που είναι σχετικά υψηλό στην Ευρώπη και μας ενδιαφέρει και στο δοκινοτικό εμπόριο αλλά και στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Οπότε θα πρέπει οι ομάδες ε, επιλογής και οι που έχουν ε, ζώα παραγωγής με υψηλό δυναμικό να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις εμπορικές συναλλαγές που θα έχουν είτε εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαλλακτικός. Ε, θα λάβω υπόψη και το θέμα των χείρων. Για τους χείρους έχουμε διαφορετική γενετική κατάσταση σε σχέση με τα βοηδή, τα εγωπρόβατα και τα υποειδή. Σε ό,τι αφορά τις ράτσες, τις φυλές, ε, προσπαθήσαμε να ορίσουμε τη φυλή, το κάνουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ορισμό, αλλιώ ε, θα υποχρεωθούμε να μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ορίσει προηγουμένως. Δεν είναι σωστό αυτό. Και υπενθυμίζω και την συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε εκτενώς πριν ε, καταφέρουμε τελικά να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Dziękuję. Σας ευχαριστούμε κύριε Νταντάν. Ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Και περνάμε στο σημείο 10, στην έκθεση του κυρίου Μέλο για τον τομέα απορροκυπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007. Είμαστε αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή για την έκθεση αυτή της πρωτοβουλίας, ενώ οι επιτροπές ανάπτυξης και ελέγχου προϋπολογισμού θα υποβάλλουν... Σήμερα θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της εκθέσεως αυτής ίδιας πρωτοβουλίας για την κατάσταση των, οργανισμών, των οργανώσεων συγγνώμη, παραγωγών καθώς και τα επιχειρησιακά ταμεία στον τομέα των ε, οποροκυπευτικών και πώς έχουν τα πράγματα μετά τη θέση εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2007. Ε, η έκθεση αυτή είναι η αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αντίστοιχη έκθεση που είχε δημοσιεύσει το Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έναν απολογισμό, μια και έχουμε ήδη κάποια χρόνια εφαρμογή τη μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ το 2007. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπήρξε μια σταδιακή βελτίωση της κατάστασης με την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ε, κυρίως αυξάνεται σταδιακά η παραγωγή που διατίθεται στην αγορά μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Και αυξάνεται και ο αριθμός των οργανώσεων παραγωγών που διαχειρίζεται επιχειρησιακά ταμεία. Βέβαια είχαμε διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό το διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαφορετική σημασία των οργανώσεων παραγωγών στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης, μεγάλες διαφορές υπάρχουν ε, μεταξύ των παλιών και των νέων ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση ΚΑΠ ε, επέφερε μερικές αλλαγές στην ειδική νομοθεσία για τα απορροκυπευτικά με την θέσπιση της κοινή οργάνωσης αγοράς ο Επίτροπος Χόγκαν κατά την ακρόασή του δήλωσε την επιθυμία του να επιφέρει κάποιες απλουστεύσεις στο καθεστώς των οροκυπευτικών ήδη κατά την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του. Θα έχουμε τώρα μια πρώτη παρουσίαση της έκθεσης από τον κύριο Μέλο και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να επανέλθουμε στο πρόβλημα, γιατί παραλαμβάνω, αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μέλο, για να μας κάνει την εισαγωγική παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι λακωνικός γιατί με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να ακούσω τους συναδέλφους. Έχουμε ε, διάφορες συστάσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της. Είναι γνωστές, δεν πρόκειται να σας κουράσω με την επανάληψή τους. Γενικώ οι περισσότερες ε, συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κατάλληλες και σωστές, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μερικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλήγει σε μια ομοιομορφία μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορές. Σε μερικές χώρες οι οργανώσεις παραγωγών ε, είναι αποτελεσματικές και έχουν ε, μακροχρόνια και ιστορική παρουσία, ενώ σε άλλες χώρες ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά και υστερούν οι οργανώσεις παραγωγών. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στο 43% το ποσοστό οργάνωσης των ε, παραγωγών. Και επαναλαμβάνω, υπήρχαν ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα σημεία φετηρή ήταν διαφορετικά. Σε ορισμένε χώρες είχαμε υψηλό επίπεδο οργάνωσης και σε άλλες πολύ χαμηλό επίπεδο οργάνωση των παραγωγών. Παρά την σταδιακή αύξηση της οργάνωσης των παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενικώ η οργάνωση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και στις περισσότερες χώρες ε, η παραγωγή των απεροκυπευτικών δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, όπως είναι η ρευστότητα, η αστάθεια των τιμών, οι κλιματικές αλλαγές ε, που θα επιδεινωθούν στο μέλλον και που αφήνουν αν μπορούσε ακόμη περισσότερο και ανυπεράσπιστους στους παραγωγούς. Οι παραγωγοί θα οργανωθούν αν πιστούν ότι με την οργάνωση αυτή θα αυξήσουν τα εισοδήματά τους και τις αποδόσεις τους. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα με οικονομίες κλίμακος και την αύξηση του οικονομικού μεριδίου των φορέων. Επίσης θα πρέπει να περιλάβουμε και το καθεστώς διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων. Να λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία και να απλουστεύσουμε το σύστημα περιορίζοντας τη γραφειοκρατία. Έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και οι διάφορες πολιτικές και εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν και την ανταγωνιστικότητα και τις τιμές. Γι' αυτό τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της κρίσης είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά την διοικητική απλούστευση του καθεστώτος. Και στα μέτρα και στις διοικητικές υποχρεώσεις των οργανώσεων παραγωγών. Θα πρέπει να αποφύγουμε το γραφειοκρατικό άχθος και την αύξηση της γραφειοκρατίας και επίση θα πρέπει να διευκολύνουμε τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών στη διενέργεια των ελέγχων. Επίσης, το θέμα της συγκέντρωσης τη εξουσία από τις μεγάλες αλυσίδε διανομής δεν είναι το αντικείμενο αυτής τη έκθεσης, γιατί εμείς έχουμε άλλη έκθεση πρωτοβουλία ε, για τις αθέμητε εμπορικέ πρακτικές, αρμόδια κατ' ουσία είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εδώ ασχολούμαστε με τον τομέα των οποροκυπευτικών, γιατί έχουμε κυρίως νοπάω οπωροκυπευτικά και σίγουρα η δυνατότητα αποθήκευση είναι πολύ πιο χαμηλή. Και αυτό αποδυναμώνει την διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών στις διαπραγματεύσεις τους με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής. αυτά και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελα να μου απαντήσει και να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Οι πληροφορίες ε, της έκθεσης ε, δεν είναι πρόσφατες. Μιλούμε για στοιχεία του 2008 με 2010. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πιο επίκαιρα και ενημερωμένα στοιχεία. Επίσης, ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, πώς πιστεύετε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το βαθμό οργάνωσης, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και τις χώρες όπου δεν υπάρχει αρκετή οργάνωση των παραγωγών. Θέλετε να προτιμάτε να δημιουργηθούν νέες ενώσεις παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες οργανώσεις. Επίσης, ε, για τη διαπραγματευτική ισχύ των οργανώσεων παραγωγών. Θεωρείτε ότι αυξάνεται με την πρότασή σας απέναντι στη συγκέντρωση των αλλιών Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διαπραγματευτική τους εσύ στην αλυσίδα παραγωγής, στην, ε, τροφική αλυσίδα. Και πώς θα ε, βελτιώσουμε την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων. Το θέμα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης είναι επίσης πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Ελπίζω να βελτιωθεί αυτή η πτυχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, άλλο σημαντικό θέμα είναι η απλούστευση. Η διοικητική απλούστευση. Δεν θεωρείτε ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό το σύστημα. Πώς θα απλουστευτεί κάπως. Θεωρείτε ότι η υπερβολική γραφειοκρατία οφείλεται στις εθνικές νομοθεσίες ή στην κοινοτική νομοθεσία. Και τέλος, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κάποια κριτήρια για την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Πιστεύω ότι χάρη στη συμβολή όλων θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέλο για την ανταλλαγή απόψε. Τώρα πρώτα ζήτησε το λόγο η κυρία Ντολαγιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαβάζοντας την έκθεση θα ήθελα να παραμείνουμε στο πλαίσιο. Στα απορροκυπευτικά τα νοπά είμαστε. Να θυμηθούμε ότι χαλάνε, δεν μπορούν να αποθηκευτούν, τα καταναλώνουμε ως έχουν, ε, με προσφορά και κατανάλωση τυχαία, διότι εξαρτάται αυτό από τις κλιματολογικές ε, συνθήκες. Ένα άλλο ιδιαίτερο σημείο, 50 διαφορετικά προϊόντα, 35 λαχανικά, 15 οπορικά. Ε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη επικοινομορφία με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ε, η λύση δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μία και μοναδική. Έχουμε μπροστά μας έναν τομέα με διαφορετικές προσδοκίες και με διαφόρους τρόπους λειτουργίας τοπική, παραγωγή, βιολογική παραγωγή, ε, μεγάλες εξαγωγές, ε, παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα κλπ. Και όλοι αυτοί οι τομείς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό εκτός κοινότητας πάρα πολύ μεγάλο. Ε, βέβαια πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη των παραγωγών και να μπορέσουν να οργανωθούν στις διάφορες αγορές που έφυξα. Η οργάνωση των ε, παραγωγών είναι ακρογωνίως ακρογωνίος Αλλά σαν παραγωγός ε, λαχανικών λέω ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες περιοριστικοί για την δημιουργία οργανώσεων παραγωγών σε αυτή την έκθεση και κάποια σημεία μου δημιουργούν απορίες, όπως το θέμα της γκρίζας οικονομίας ε, που αφορά τους μη οργανωμένους παραγωγούς και δημιουργεί προβλήματα. Συμφωνώ με τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των παραγωγών, ο κίνδυνος ε, απώλειας των κρατικών ενισχύσεων επίσης που αναφέρεται στην, ε, στην έκθεση αυτή αλλά οι, οι οργανώσεις της αγοράς δεν είναι η αποκλειστική λύση. Ε, παραμένει όμως ακρογωνίως λίθος ε, του, της όλης προσέγγισης. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις που είναι σε ηγετική θέση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει η ανάγκη να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των αγορών ανεξάρτητα από το μέγεθος που έχουν οι δομές Λέγεται ότι καλό μέγεθος είναι αυτό που ε, αφήνει να πατάει κανείς με το πόδι στο έδαφος. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα απορροκυπευτικά. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη δύναμη των παραγωγών, να διευκολύνουμε την, ε, την συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών, αλλά να συμμετέχουν και ανεξάρτητοι παραγωγοί, διότι στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια υπάρχουν και μεγάλοι ανεξάρτητοι φορείς και αν θέλουμε να προβλέψουμε και να διαχειριστούμε τις κρίσεις και να προωθήσουμε τα προϊόντα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να συμμετέχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς. Όσον αφορά τα συμπεράσματα της ε, εκθέσεως, κάτι που ανέφερε και ο συνάδελφός μας μέλο προλίγου, είμαστε στην περίοδος 2008-2010, τέλος 2014, ε, ξεκινήσαμε, είμαστε 2014, έγιναν πολλά, χρειάζεται επικαιροποίηση λοιπόν των μέτρων όσον αφορά ε, τους χρειάζονται επιχειρησιακά προγράμματα για να διευκολύνουν τα προγράμματα των οργανώσεων και έτσι να διευκολύνουμε την ενίσχυση την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών ε, περισσότερο από την τιμή των προϊόντων χρησιμοποιώντα λοιπόν ε, να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής ε, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα διάθεση των προϊόντων σε καλύτερες τιμές τώρα ε, και το θέμα του ανταγωνισμού, το δικαίωμα του ανταγωνισμού δεν αφαιρείται στην έκθεση. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να συνδέσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με την αναθεώρηση που θα γίνει και στην αναγνώριση των οργανώσεων των παραγωγών και στη δυνατότητα να υπάρχει συνεργασία και με τους ανεξάρτητους ευρωπαίους παραγωγούς σε ευρύτερη κλιμάκα θα πρέπει να μην εξετάζουμε το θέμα μόνο από μακροοικονομική σκοπιά, αλλά και από μικροοικονομική, διότι εκεί βρίσκονται και ενδεδειγμένε λύσει. Τέλος, έχω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Διότι ίσω υπάρχουν κάποιες διέξοδοι. Ε, μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το εύρο ε, των προτάσεων, την εμβέλεια των προτάσεων που σκέφτεται να μα υποβάλει. Σας ευχαριστώ κύριε Σερντός. Φυσικά όλοι κατανόησαν ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων των παραγωγών στις χώρες αυτές. Ακούσαμε επίσης να ε, τίθεται και το ερώτημα. Ποιος είναι ο στόχος, ήταν το ερώτημα. Ποιος είναι ο στόχος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε την όλη κατάσταση, όλους τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα αναλύσει εκ νέου τα στοιχεία Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν οι επιδοτήσεις, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τις οργανώσεις των παραγωγών. Δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα, πρέπει να πλουστεύσουμε το σύστημα, το γνωρίζουμε όλοι. Κάθε μέρα λέμε ότι πρέπει να πλουστεύσουμε τις διάφορες διαργασίες και κυρίως στα πλαίσια των οργανώσεων των παραγωγών. Πιστεύω προσωπικά και είναι η άποψή μου αυτή, ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλα τα ζητήματα, να τα επαναπροσεγγίσουμε και θα πρέπει να ξανατεθεί το ερώτημα ποιος είναι ο στόχος. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Στόχος είναι να έχουμε όλο και περισσότερες οργανώσεις παραγωγών. Αυτό είναι ο στόχος. Ευχαριστώ. Ε, grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπε και συνάδελφος που προηγήθηκε. Θα πρέπει να εστιαστούμε στον τομέα αυτό για να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν οι οργανώσεις των παραγωγών. Και εγώ σημείωσα, όπως και ο εισηγητής, κάποια προβληματάκια όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω ότι αυτές τις εβδομάδες θα καταφέρουμε να εξηχνιάσουμε τα διάφορα θέματα. Ε, πάση περιπτώσει, όταν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και τα στοιχεία που διαθέτουμε. Τώρα, ε, όσον αφορά η οργάνωση στον απορροκυπιστικό τομέα δεν είναι πάρα πολύ καλή, δεν είναι πολύ καλά οργανωμένη η παραγωγή. Υπάρχει χαμηλό επίπεδο. Ε, οι μικρές διαστάσεις των οργανώσεων, περιορισμένη κάλυψη κάποιων οπορικεπιστικών προϊόντων από πλευράς των οργανώσεων των παραγωγών και η έλλειψη διαχείρισης επαγγελματικής ίσως είναι βασικά αδύναμα σημεία του τομέα. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ανισορροπίες περιφερειακές όσον αφορά την οργάνωση των παραγωγών των οποροκυπευτικών. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να την ανάπτυξη των οργανώσεων αυτών σε κάποιες περιφέρειες και μεταξύ των κρατών μελών. Βασικό πρόβλημα είναι ο περίπλοκος χαρακτήρας των ε, διαδικασιών που ε, προβλέπονται για την αναγνώριση των ε, οργανώσεων. Αυτά είναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί όπως και για τη δημιουργία και τη διαχείριση και τη δημιουργία οργάνωσης αναγνωρισμένης ε, απορροκευτικών προϊόντων είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία και έτσι υπονομεύει ε, ίσως και τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει η μεταρρύθμιση. Άλλοι κανόνες του καθεστώτος είναι περίπλοκοι για, τους, ε, για τις οργανώσεις περιοχών. Το θέμα αποδοχής διαφορών ειδών, η παροχή διαφόρων τεχνικών μέσων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε κάποια κράτη-μέλη να δώσουν οικονομική ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο στι οργανώσει των παραγωγών που λειτουργούν σε περιφέρειε όπου το επίπεδο των οργανώσεων των παραγωγών στον προκυπτικό τομέα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Δυστυχώ μόνο έξι χώρε ε, καλύπτονται από αυτό το μέσο και η μεταρρύθμιση του 2007 του τομέα των απορροκυπευτικών δημιούργησε και διάφορα εργαλεία διαχείρισης και πρόληψης των κρίσεων στα, στα επιχειρησιακά προγράμματα της οργανώσης των παραγωγών, όπως η υποστήριξη εκτός ε, των ε, αγορών. Η προσφυγή σε αυτά τα εργαλεία ήταν πάρα πολύ περιορισμένη παρά την κρίση που ε, έπληξε την αγορά. Σε κάποια κράτη-μέλη τα προγράμματα τα επιχειρησιακά αποτελούν ένα μέσο που χρησιμοποιείται ελάχιστα ή καθόλου για την αύξηση της εμπορικής αξίας ε, των ε, προϊόντων που ιδρύεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις των παραγωγών για να προωθήσουν τη συγκέντρωση της προσφοράς. Αυτό οφείλεται στην αιμονή, στη μικρή συμβασιακή ε, δύναμη που έχουν οι οργανώσεις περιεχών, ε, συγγνώμη, παραγωγών. Ε, και είναι πολύ λίγες οι οργανώσεις των παραγωγών για να συνάψουν συμφωνίες και μικρή διάστασή τους και γι' αυτό. θα πρέπει λοιπόν να ακολουθηθεί η σωστή διαδρομή ούτω ώστε να ενισχύσουμε τι οργανώσει των παραγωγών και ταυτόχρονα, όπω έλεγε ο προλαλή σα συνάδελφο, θέλουμε να συνοδεύσουμε και τους παραγωγούς, του. ανεξάρτητους, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε επεξεργαζόμενοι κάποια συγκεκριμένα σημεία, τα οποία ήθελα να συνοψίσω. Κυρίως να πούμε σαφώς ποιοι είναι οι στόχοι, οι προτεραιότητες και να εξηγήσουμε σαφώς ε, ποσοτικά τους στόχους. Μόνο έτσι θα είναι δυνατό να προσμετρήσουμε άμεσα και αντικειμενικά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να κατευθύνουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα προς την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων που συνάδουν με τον στόχο της βελτίωσης παροχής και της ανταγωνιστικότητας ε, της συνολικής του συστήματος τοποκυρπιστικού. Και θα είναι πιο εύκολο να ακολουθήσουμε τη δραστηριότητα αξιολογήσεως των εθνικών στρατηγικών στο σύνολό τους και να έχουμε σωστές διορθωτικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα αποκλίνουν από τους αρχικούς σκοπούς των σχεδίων. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε σε σχέση με το παρελθόν τη δράση συμπράξεων με τους βασικούς φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και που διαχειρίζονται τα επιχειρησιακά προγράμματα, τόσο ώστε να προσανατολίσουμε καλύτερα τι επιλογέ όσον αφορά στρατηγικέ απαιτήσει του τομέα. Τρίτο σημείο, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στενότερο συντονισμό με τα άλλα μέσα προγραμματισμού εθνικού και περιφερειακού. Τέταρτο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε του ε, κανόνε ευρωπαϊκού, ούτω ώστε να δώσουμε νέα προώθηση διαδικασία τη ομοδοποίηση, ε, ανεβάζοντα τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων και θα πρέπει να υπάρχει το σύστημα να είναι και θα πρέπει τα κοινοτικά προγράμματα να οδηγήσουν σε καινοτόμα μέσα. Οπότε μια σύμπραξη ευρωπαϊκή για καινοτομία. Όλα αυτά ακολουθούν την κατεύθυνση της απλούτευσης ε, των διαδικασιών για έναν τομέα ε, που χρειάζεται υποστήριξη της κυβερνήσεως και τελικά οι κυβερνήσεις να, μην, ε, να διευκολύνουν την όλη κατάσταση και όχι να, να δημιουργούν περισσότερα, στενότερα πλαίσια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά πράγματα ήδη υπόθηκαν από τους διάφορους ε, ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλο καταρχάς για την ε, ποιότητα της εκθέσεώς του. Ο τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, το γνωρίζουμε στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα και από την ε, ισχύουσα μεταρρύθμιση ε, λίγα πράγματα άλλαξαν όσον αφορά τις ε, παρεμβάσεις και ελάχιστα άλλαξαν όσον αφορά το καθεστώς των απορροκεπιστικών προϊόντων. Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Υπάρχουν ανεπάρκειες όσον αφορά την υποστήριξη στον τομέα των απορροκεπιστικών προϊόντων και αναφέρθηκε προηγουμένως διότι πολλοί παραγωγοί δεν την χάνουν υποστήριξης. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι το αίτημα που πολλοί ανέφεραν την, ε, χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων. Δεν μπορούμε να εργαστούμε σοβαρά το 2014 με πληροφορίες που ε, είναι πολύ επιρχιωμένες. Είναι βασικό στοιχείο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία και τον πολύπλοκο χαρακτήρα του θέματος. Βλέπουμε ότι λόγω ελλείψεως οργανώσεων επαγγελματικών των παραγωγών, όπως υπογραμμίστηκε και είναι πολύ μικρές οι οργανώσεις, η παραγωγή πολύ μικρή είναι αυτοί που πλήττονται. Και έχουν και πολύ μικρή διαπραγματευτική δύναμη έτσι. Και εντό του τομέα. Όταν βλέπουμε τις ενισχύσεις που χορηγούνται, οι πιο μεγάλες οργανώσεις των παραγωγών, όταν υπάρχουν αυτές, αυτές λαμβάνουν ε, τη μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση της ε, Ένωσης. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αληθεύει, όπως υπόθηκε, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε, τις, να στηρίξουμε τη σχέση μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων των παραγωγών και το άλλο που θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν την ελκυστικότητα των οργανώσεων των παραγωγών, αυτό είναι ένα σημείο βασικό, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε την ε, ανάπτυξη, την αύξηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων. Ο κ. Καπούτο αναφέρθηκε σε αυτό επίσης, στο θέμα της βελτιώσεως των μέσων που έχουμε για τη διαχείριση και πρόληψη των κρίσεων. Εκεί υπάρχουν πραγματικές προτάσεις που μπορούν να γίνουν και περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες προτάσεις πολύ ακριβέστερες και συγκεκριμένε σε αυτό το θέμα. Γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα των τιμών. Και τέλος κάτι άλλο που αναφέρθηκε, το θέμα της απλουστεύσεως του όλου μηχανισμού που υπάρχει. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος ε, ε, το τόνισε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, αλλά να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για να απλουστεύσουμε πραγματικά ε, τον όλο μηχανισμό, αν θέλουμε να επιτρέψουμε να υπάρξει βελτίωση της καταστάσεως τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Είναι όντως κάπως ε, απερχιωμένη η έκθεση, αλλά στην πρώτη σελίδα είναι... υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Υπάρχει σημαντική διαπίστωση της μείωσης ε, της ε, ευρωπαϊκής παραγωγής απορροκυπευτικών στην περίοδο αναφοράς. Είναι πραγματικά λυπηρή αυτή η διαπίστωση, γιατί η περίοδος 2007-2010 είναι μια περίοδος σχετικής οικονομικής ευμάρειας ε, και μεγάλης αγοραστικής δύναμης. Και ξέρουμε ότι τα παρακυβευτικά είναι από τα προϊόντα που βελτιώνουν τη διατροφή και υπήρχε δυνατότητα ε, αγοράς. Αν τότε όμως δεν καταφέραμε να καλύψουμε την, ε, ούτε την εσωτερική ζήτηση, ούτε κερδίσαμε σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές. Ενώ αυτές ήταν βασικές μας προτεραιότητες και στόχοι κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η μεταρρύθμιση του 2007 δεν τροποποίησε ριζικά τις ισορροπίες. Όσοι ήταν καλά οργανωμένοι παραμένουν, όσοι δεν ήταν καλά οργανωμένοι δεν βελτιώθηκαν. Ούτε μπόρεσαν να λύσουν κάποια προβλήματα με τα μέσα που προβλέψαμε. Γιατί πόσα μικρές πώς, μικρέ οργανώσει μικρές οργανώσεις παραγωγών μάλλον θα κάνουν πρόληψη και διαχείριση κρίσεων. Για να έχει κάποιος βάρος σε μια κρίση θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη δράση και αποφασιστική. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο από μικρές οργανώσεις παραγωγών. Επίσης, στην έκθεσή μας για την κοινή οργάνωση αγοράς ζητήσαμε να θεσπιστούν κάποιες διατάξεις για να βελτιωθεί το η εμβέλεια των οργανώσεων παραγωγών ε, για να συσπηρωθούν σε πολύ μεγαλύτερες οργανώσεις η παραγωγή και να έχουν μεγαλύτερο βάρος στις εξελίξεις και επίσης ζητήσαμε απλούστευση κάποιων μηχανισμών παρέμβασης. Η νέα πολιτική δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ακόμη γιατί περιμένουμε ακόμη τα σχετικά κείμενα. Πριν από ένα χρόνο τροποποίησαμε την κοινή οργάνωση αγοράς Βρισκόμαστε ήδη στη μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης, ενώ δεν μπορέσαμε καν να κάνουμε έναν απολογισμό της πρώτης μεταρρύθμισης και το α, κατά πόσο ήταν αυτή η αποφέλης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ροπέ. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai ačiū pranešėjui už pranešimą. Manau, kad klausimas pakankamai įdomus ir tai, kad e, Ευχαριστώ. Το θέμα της έκθεσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Μετά το 2007 που άρχισε η μεταρρύθμιση δεν αλλάξαν πολύ τα πράγματα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ίσως δεν χρειαζόταν ή δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Το 43% των... Ε, είναι παραγωγή Πολλές φορές δεν υπάρχουν οργανώσεις παραγωγών. Προσπάθησα να εμπαθύνω στο αίτιο γιατί μου φαίνεται ότι έχουν προοπτικές και είναι χρήσιμες οι οργανώσεις παραγωγών. Όταν όμως μιλήσουμε σε ενώσεις παραγωγών, βλέπουμε ότι δεν θέλουν νέα μέλη. Ίσως θα έπρεπε να ενισχύσουμε περισσότερο αυτές τις οργανώσεις παραγωγών για να γίνουν δεκτά και νέα μέλη. Τώρα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι μεγάλες οργανώσεις δεν παίρνουν νέα μέλη και οι μικρές οργανώσεις δεν έχουν δυνατότητες οι, μικροί παραγωγοί δεν μπορούν να συστήσουν οργάνωση παραγωγών. Οι οργανώσεις παραγωγών που υπάρχουν δεν έχουν λόγο να, πάρουν, να δεχθούν νέα μέλη. Γιατί ήδη έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς και έχουν πολύ καλές προοπτικές. Σε σχέση με διαπραγματευτική ικανότητα, κέντρα πώλησης, ε, αγορές. Οπότε είναι εξασφαλισμένη, εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγωγής τους. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Για να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε νέα μέλη για τις οργανώσεις των παραγωγών. Και να έχουμε αισθητά αποτελέσματα. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε ενδεχομένως συγκεκριμένα μέτρα που θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των οργανώσεων παραγωγών να δεχτούν νέα μέλη. Το σύστημα των οργανώσεων παραγωγών ε, θα έπρεπε γι' αυτό να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη και να προσαρμόζεται σε αυτές γιατί και η γεωργία και το περιβάλλον διαφέρουν στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την αρνητική γενικότερη διάθεση που αναφέρεται εδώ δεν τη συμμερίζομαι οι οργανώσεις των παραγωγών. Είναι προαιρετική προσφορά που δημιουργήσαμε και το διαθέσαμε στους παραγωγούς οπωροκυπευτικών και νομίζω ότι έχουν ίδια ευθύνη παραγωγή να χρησιμοποιήσουν ή όχι το μέσον αυτό. Λέμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν προχώρησε η συνεργασία. Για να δούμε γιατί συνέβη αυτό επειδή δεν λειτουργήσε το εργαλείο μας, δεν λειτουργήσε η νομοθεσία ή μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι. Σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιφέρειες της Ένωσης μπορεί να μην υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας και οι παραγωγοί να μην θέλουν να συνεργάζονται και να συνασπιστούν. Εγώ είμαι από μια περιφέρεια όπου το παράγεται το 15% 3,5 δις κιλά μήλα το 2007 τα μήλα αυτά επολούνται από 40 εμπόρους. Τώρα είναι δύο γιατί λειτουργήσε η συνεργασία. Αν δεν υπήρχε συνένωση παραγωγών δεν θα έχει συνέβαινε κάτι τέτοιο και τώρα έχουν και καλή θέση στην αγορά εναντί των μεγάλων ε, παραγόντων στην αγορά. Σούπερ μάρκετ και το θέλουμε αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι οι παρεμβάσεις μας είναι υπερβολικά λίγες. Αυτό δεν είναι δουλειά των οργανώσεων παραγωγών, δεν είναι δηλαδή να παίρνουν τα προϊόντα από την αγορά, αλλά να θέτουν προϊόντα στην αγορά και η παρέμβαση θα πρέπει να είναι μια εξαιρετική κατάσταση. Ε, όχι ο κανόνας, θα είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι να υπάρχουν οργανώσεις που στις ε, μεγάλες αλυσίδες θα πολλούν προκυπευτικά, όχι να αποσύρουν προϊόντα από την αγορά. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το μέσον αυτό, να το σκεφτούμε. Όχι όμως ε, τα κριτήρια πρόσβασης να τα ε, υποβαθμίσουμε για να μπορεί να γίνεται ή μάλλον όχι να μην μπαίνει ο καθένας, βεβαίως ο καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπει, αλλά να είναι τόσο μικρές οι οργανώσεις ε, παραγωγών ε, για να αυξάνουν ε, αναγκαστικά τα μέλη. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετούνται οι γεωργοί έτσι. Και, όπως είπα, να ρωτήσουμε, όπου δεν λειτουργήσε το σύστημα και είναι οργανωμένοι μόνο η μισή και η άλλη μισή όχι, ε, θα πρέπει να δούμε γιατί και στη δική μου χώρα ε, σε ορισμένες περιφέρειες δεν λειτουργήσε το σύστημα αλλά πρέπει να δούμε επειδή δεν το θέλουν οι αγρότες ή επειδή δεν εξυπηρετεί. Ευχαριστώ κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος Μέλο, Η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στηρίχθηκε σε πληροφορίες και δεδομένα των κρατών μελών για την ε, εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Καθεστώτος Απορροκυβευτικών και με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνουν και τις εκθέσει τους. Όπως ξέρουμε, η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν θα αλλάξει ριζικά τον καθεστώς των απορροκυπευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια και η κοινοτική ενίσχυση προσφέρεται στις οργανώσεις παραγωγών μόνο μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με δύο μόνο εξαιρέσεις, τις ενώσεις παραγωγών που ιδρύουν επιχειρησιακό ταμείο με συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων. Αυτές είναι οι δύο εξαιρέσεις. Και πιστεύω ότι είναι σωστή αυτή η έμφαση που δίνουμε στις ε, οργανώσεις παραγωγών, γιατί έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ και μια πιο στεντόρια φωνή στις διαπραγματεύσεις, αλλά μην ξεχνούμε ότι σε μερικές χώρες δεν είναι τόσο καλά οργανωμένη η παραγωγή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τον ίδιο τρόπο χώρες που έχουν ε, ισχυρά οργανωμένους παραγωγούς στα προκυπευτικά και χώρες που στερούνται τέτοιου επίπεδου οργάνωσης και που είτε είναι αδύναμες οργανώσεις παραγωγών είτε δεν υπάρχουν. Αλλιώς ε, θα επικεντρωθούμε μόνο στην ε, κατάσταση που ισχύει σε ορισμένες χώρες και δεν θα καλύψουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ και εγώ ήθελα να υπογραμμίσω πολύ σύντομα αυτό που ο συνάδελφος Ντόρφμαν είπε προλίγου. Συζητάμε ένα μέσο αυτό το θέμα και των απορροκυπευτικών είναι ελάχιστε οργανώσει που έχουμε. Είναι τα ελάχιστα μέσα που έχουμε στην αγροτική πολιτική στην Ευρώπη που ευνοεί η βελτίωση τη οργανώσεω των επιχειρήσεων και των παραγωγών στον τομέα, κυρίω των μικρών παραγωγών. Είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί διότι αναμφισβήτητα υπήρξε μια βελτίωση ε, η οργάνωση ήταν κατακαιρματισμένη. Είχαμε από πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελάχιστες μιλάμε για προκυπευτικά ε, προϊόντα με δυσκολίες οργανωτικές και καταφέσαμε μέσω συνεταιρισμών ή οργανώσεις παραγωγών να τις συναθρήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αγορά ε, που είναι πολύ πιο καλά οργανωμένη. Όσον αφορά ε, ε, η λειτουργία κάποιων αποτελεσματικότητα κάποιων μέτρων για την κρίση των αγορών δεν πέτυχαν διότι όταν κάνουμε τα ρύθμιση του 2007 δεν δώσαμε επαρκή ευελιξία ε, στις οργανώσεις των παραγωγών για να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Φέτος με την κρίση που διαπιστώσαμε με το εμπάργκο το ρωσικό πώς θα μπορούσαμε να, να βοηθήσουμε τις οργανώσεις των παραγωγών, να επιτρέψουμε μια πόση από την αγορά. Είδαμε μια έκρηξη των μέσων για την κρίση της αγοράς. Θα το βλέπαμε αυτό αν μπορούσαμε τελικά να επιτρέψουμε στις οργανώσεις των παραγωγών να κάνουν τις αποσύρσεις. Θέλαμε να ενισχύσουμε και να κάνουμε πιο ανταγωνιστικούς ε, τους ε, παραγωγούς. Λειτουργούν εργάσεις των παραγωγών. Μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε αυτά, ναι, σίγουρα. Αλλά είναι και ένα ερώτημα που επιθύνω προ τον εαυτό μου και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε είναι οι ιδέε για να τι κάνουμε πιο ανταγωνιστικέ οργανώσει αυτέ. Εγώ δεν θα ήθελα αυτές οι υπερβολές μεταρρυθμιστικές να οδηγήσουν σε μια επιδίνωση. Αυτό που ζητούσε και ο κύριος ε, Μέλο, διότι εξετίμησα τόσα μας είπε στην ε, παρέμβασή του κύριος Μέλο. Κύριε κυρία Πετήρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, συνάδελφο Μέλο για την έκθεση που ετοίμασε και την εισαγωγή που μας έκανε. Πολύ εύστοχα ε, παρουσίασε τα προβλήματα των κρατών μελών και ελπίζω να δώσει απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις του κυρίου Μέλλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί εστερνίζομαι και εγώ αυτές τις απορίες ε, και ασχολούμαι κυρίως ε, για, τις, για τους μικρούς παραγωγούς. Έχουμε μόνο 43 μεγάλες ομάδες οργανώσεις παραγωγών. Είναι ανησυχητικό αυτό το στοιχείο, ελάχιστη οργάνωση, πολύ μικρή στήριξη. Φαίνεται ότι τα μέτρα που θεσπίσαμε δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί κατά πόσο θα πρέπει να αναθεωρήσει το πρόγραμμα προκειμένου να δώσει περισσότερα κίνητρα στους παραγωγούς για να οργανωθούν σε οργανώσεις παραγωγών για να αυξήσουν και την διαπραγματευτική τους ισχύ στην αγορά και στις διαπραγματεύσεις με τις αλυσίδες διανομής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Περόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τη Μολδαβία αν θα, θα, θα δεχόταν αγορά στα απορροκυπευτικά μας. Το καθεστώς των απορροκυπευτικών που υιοθετήθηκε το 2007 καταδικάζει αυτή την κρίση σε μια έναη κρίση. Χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία για τη ρύθμιση. Η, η οργάνωση των παραγωγών, στις οργανώσεις των παραγωγών δεν μετράει ε, σε τίποτα όσον αφορά τα μεγάλα κέντρα αγορών, ε, ούτε στον αθέμητο ανταγωνισμό των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Χειρότερα, το κοινωνικό dumping μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όλος είναι ιδιαίτερα καταστροφική για αυτή αυτό τομέα που ζητά πάρα πολλά εργατικά χέρια αυτό το κοινωνικό dumping ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί σαν ισορροπίε, διότι επιτρέπει στα κέντρα αγορά των μεγάλων εταιριών να ασκούν πιέσει και να πιέζουν τι τιμέ προ τα κάτω στι διαπραγματεύσει για τη σύναψη συμβάσεων. Για του Γάλλου παραγωγού ε, που έχουν εργατικό κόστος ε, τρεις φορές πιο ψηλότερο από ό,τι έχουν Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί η κατάσταση για μα είναι αφόρητη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μέλο για τη σημερινή του παρέμβαση, την παρουσίαση. Θέλω να επικρίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να πω ξεκάθαρα το εξή. Γιατί εργαζόμαστε με ε, στοιχεία. Σίγουρα έχουν πιο επικαιροποιημένα στοιχεία από αυτά του 2010. Θέλουμε να ξέρουμε πού είμαστε τώρα, όχι πού βρισκόμασταν το 2010. Ε, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει εναλλακτικέ αγορές υπό το φως του ρωσικού εμπάργου αλλά όχι μόνο αυτό θα πρέπει να εξετάσει και το θέμα της αγοράς του γάλακτος όταν απαλλαχθούμε από τις ποσοστώσεις του γάλακτος. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει λύσεις. Θέλουμε περισσότερες τέτοιες οργανώσεις παραγωγών. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε τους παραγωγούς να δημιουργήσουν οργανώσεις. Μπορούμε να τους δώσουμε κίνητρα όμως. Ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιωθεί το επίπεδο οργάνωσής τους. Αυτό ισχύει για τους μικρούς ε, παραγωγούς αλλά και για τους μεγάλους παραγωγούς. Πρέπει να μπορούν να ε, αντιμετωπίσουν την κρίση που την εμπνέει η Ρωσία και θα έπρεπε να μπορούν να οργανώνονται και μεταξύ τους καλύτερα. Να οργανώνονται οι ίδιοι καλύτερα. Η μικρή παραγωγή θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού ε, μηχανήματα και θα πρέπει επίσης να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που ασκούν πάνω τους τα σούπερ μάρκετ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα, διότι για την ώρα δεν ξέρω τι μπορεί να μας φέρει το μέλλον. Ο κύριος Σεμπαστιά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να σε συγχαρώ τον κύριο Μέλο για το έργο του, για την έκθεσή του. Επισήμανε ένα πρόβλημα τα παροχημένα στοιχεία. Ε, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου, έχουμε παράδοση ε, οργανώσεων παραγωγών. Παράγουμε πορτοκάλια, ελαιόλαδο, σημαντικά προϊόντα για την Ευρώπη. Στόχος των οργανώσεων παραγωγών είναι να προστατεύσουν κυρίως τους μικροπαραγωγούς, και να βοηθήσουν τη διάθεση σε εμπορία, τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του. και φυσικά να βοηθήσει και τι επενδύσεις που είναι σημαντικό για τη βελτίωση τη παραγωγής. Ακόμη όμως και σε αυτές τις οργανώσει παραγωγών έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με τη διάθεση στην αγορά ε, των ε, προϊόντων. Το πρόβλημα προέρχεται από, την, από τον αθέμητο ανταγωνισμό με τα προϊόντα τρίτων χωρών. Και εδώ δεν φταίνε οι οργανώσει των παραγωγών, αλλά οι ευκολίες που έχουν τρίτες χώρες και οι σχετικά χαλαρές προδιαγραφές είτε ποιοτικές είτε κοινωνικές κάτι που δημιουργούν τον ανταγωνισμό με τους Ευρωπαίους γεωργούς που πρέπει να πληρούν πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Το θέμα δεν είναι λοιπόν οι οργανώσεις των παραγωγών, αλλά ο θέμητος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Εράς, Εράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τέσσερις προτάσεις που μας έκανε πέρυσι για τα τέσσερα πιθανά σενάρια ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν μη τι άλλο αναγνώρισε την αναποτελεσματικότητα των εφισταμένων ε, μηχανισμών διαχείρισης της κρίσης και τις διοικητικές δυσκολίες ό,τι αφορά τη διαχείριση των επιχειρησιακών ταμείων ε, από πλευράς οργανώσεων παραγωγών στα απορροκυπευτικά. Αυτό θα πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα στο μέλλον και πολύ σωστά το επισήμανε από την αρχή ο κύριος Μέλο γιατί γνωρίζει την κατάσταση, μια και κατάγεται από μια χώρα που είναι σημαντική χώρα απορροκυπευτικών. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία στο Συμβούλιο ε, εντόπισαν με σαφήνεια και εύστοχα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στου μηχανισμού πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων και για το ύψο των αποσύρσεων, αλλά και για την επικαιροποίηση των ε, ενισχύσεων για τις αποσύρσεις. Επίσης θα πρέπει να γενικεύσουμε την δωρεάν διανομή μεταποιημένων προϊόντων και να προβλέψουμε και κάποια νέα μέσα διαχείρισης. Κάποιες ασφάλειες, αμοιβεοποίηση και γενικώ ενημέρωση, επικαιροποίηση κάποιων μηχανισμών που ισχύουν για τα παρακυβευτικά. Επίσης, το παρατηρητήριο των τιμών, κάτι που μας λείπει. Αν δεν θεσπίσουμε παρατηρητήριο των τιμών που θα παρακολουθεί τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ελέγχει τις ποιότητες που παράγονται, που διατίθεται στην αγορά και την προσαρμοστικότητα του τομέα να καλύψει τη ζήτηση, δεν θα έχουμε πραγματικές και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο παρατηρητήριο των τιμών. Το ίδιο είπαμε και για την τροφική αλυσίδα. Χρειαζόμαστε και στην περίπτωση αυτή το παρατηρητήριο των τιμών. Κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να επισημάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο νέος μηχανισμός σοβαρών κρίσεων. Δεν είναι μία επιπλέον δαπάνη. Απλώς θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια των οργανώσεων παραγωγών για ένα σύστημα ε, που προβλέπει ε, αντιμετώπιση της κρίσης, ιδιαίτερα μια σοβαρή κρίση για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Αυτός ο μηχανισμός σοβαρών κρίσεων και διαχείριση σοβαρών κρίσεων θα ήταν πολύ αποτελεσματικός και θα βοηθούσε πολύ και τις οργανώσεις παραγωγών αλλά και τους ανοργάνωτους παραγωγούς. Γιατί όπως είπε ο Επίτροπος Τσόλος στην προηγούμενη Επιτροπή, είναι το γεγονός ότι οι παραγωγοί δεν θεωρούν ε, ωφέλιμο το να προσχωρήσουν σε μια οργάνωση παραγωγών. Θα πρέπει λοιπόν να τους δείξουμε ότι είναι ελκυστική η συμμετοχή σε μια οργάνωση παραγωγών, όχι μόνο σε περιπτώσεις παχιών αγελάδων, αλλά και σε περιπτώσεις συχνών αγελάδων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης. Ελπίζω στο σχέδιο νέας κοινής οργάνωσης αγοράς που θα μας στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη νέα πραγματικότητα και τις νέες ανάγκες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Διευθυντής, ο κύριος Κολτέ. Θα ήθελα να σας ε, επισημάνω ότι λίγο πριν τις 5 πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί στις 5 θα έρθει ο Επίτροπος Χόγκαν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Να πω καταρχήν ότι χαιρετίζουμε ε, ιδιαίτερα την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του κυρίου Μέλου και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί του πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα μετά την έκθεσή μας του Μαρτίου. Πολύ σύντομα να βάλω την έκθεσή μας, να βάλω ένα πλαίσιο. Η έκθεσή μας αντιμετωπίζει τρεις βασικές προκλήσεις στον τομέα των οποροκυπευτικών που εντοπίστηκαν και από τους ε, ευρωβουλευτές. Πρώτον, μείωση κατανάλωση οποροκυπευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ανάγκη για αυξημένη και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των παραγωγών, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί εναντί τρίτων χωρών και εισαγωγή. Και, όπως είπαν πολύ, απόψε, για να ενισχυθεί η θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού η τρίτη πρόκληση είναι πώς θα γίνεται η διαχείριση κρίσεων στον τομέα των οποροκυπευτικών. Που αυτό διαφέρει βέβαια πολύ από τις άλλες αγορές γιατί είναι βαλίωτα τα προϊόντα αυτά και οι αγορές είναι πολύ ανελαστικές. Και αυτά τα δύο στοιχεία είναι αντικειμενικά, δεν αλλάζουν, ούτε η Κομισιόν δεν μπορεί να τα αλλάξει. Και αυτό σημαίνει και σήμαινε πάντα ότι ο τρόπος διαχείρισης των αγορών οποροκυπευτικών είναι διαφορετικό από το γαλακτοκομικό ή το τομέα του βοηού κρέατος ή το τομέα των ε, δημητριακών. Είναι άλλος τομέας που θέλει διαφορετική προσέγγιση. Πάντα ήταν αυτή μια αγορά που ήταν αρκετά ανοιχτή και φιλελεύθερη για να το πω έτσι και το μόνο μέσο που έχουμε εκτός από την προστασία στα σύνορα για να εμποδίζουμε τις φθηνές εισαγωγές είναι η οργανώση των παραγωγών. Αυτό που λέμε σε αυτή την έκθεση του Μαρτίου είναι ότι είμαστε πολύ απογοητευμένοι όπως και εσείς σχετικά με την αύξηση του ποσοστού οργάνωσης των παραγωγών. Είναι απογοητευτικό το χαμηλό ποσοστό, πάντως υπάρχει αύξηση. Και αν δούμε τα νούμερα, το 2000, ε, από το 2007 εκεί ήταν 37% το ποσοστό των παραγωγών που ήταν οργανωμένη σε οργάνωση παραγωγών και το 2010 ανέβηκε στο 43. Το 37 στα 43 λοιπόν. Πρόοδος, αλλά βραδία και ανεπαρκής. Και θα διαθέσω στη γραμματεία της Επιτροπής τα πρόσφατα στοιχεία, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά είναι λίγο παλιά στοιχεία και είμαι βέβαιος ότι έχουμε από το 2011 στοιχεία ήδη. Πολύ σύντομα θα πάρουμε και από το 12 τα ποσοστά. Αλλά γεγονός είναι ότι ε, περιμένουμε από τα κράτη-μέλη τα στοιχεία αυτά. Δεν τα έχει η ίδια η Κομισιόν. Πρέπει να τα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μα τα δώσουν και υπάρχουν, υπάρχει καθυστέρηση. Πρόοδο, ναι, λοιπόν, αλλά όχι αρκετή. Έτσι υπάρχουν μείζονες προκλήσεις που παραμένουν και είναι εντυπωσιακό αν δείτε τα στοιχεία ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπως η δική μου χώρα όπου η οργάνωση είναι σχεδόν 100% στην Ολλανδία. Ενώ ιδιαίτερα σε κάποια νέα κράτη-μέλη είναι μηδενική σχεδόν είναι η οργάνωση. Αυτό είναι ατυχές και ιδιαίτερα ανησυχητικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό μεταξύ άλλων έγινε η έκθεση και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητάμε μαζί σας το θέμα αυτό και με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι θα κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δύο πράγματα μπορώ να αναφέρω ήδη, ότι ο Επιτροπός μου, ο Επίτροπος Χόγκαν ήδη έχει δεσμευτεί εδώ στην Ακρόαση όταν ήρθε για να κάνει ε, επανεξέταση και αναθεώρηση των δυνατοτήτων απλούστευση στον τομέα και δεύτερον η Κομισιόν δεσμεύτηκε ε, υπέρ μιας μεταρρύθμισης ολόκληρου του καθεστώτος οποροκυπευτικών το αργότερο το 2018. Οπότε αυτά είναι τα δύο σημεία που έχουν ήδη ξεκινήσει και την απλούστευση την ξεκινήσαμε και την πιο θεμελιώδη μεταρρύθμιση που ε, ε, συμπεριλαμβάνει ε, τροποποίηση της νέας πράξης μπορεί να γίνει το 2018 ή και νωρίτερα. Και εδώ η έκθεση του κυρίου Μέλο είναι πολύτιμη συμβολή στη διαδικασία. Να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις ταχιστά τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση της ελλειπούς οργάνωσης σε πολλά κράτη-μέλη των παραγωγών. Αυτό που κάνουμε ήδη είναι να επιδοτούμε μέχρι 4,1% της αξίας το, της παραγωγής που πάει στην εμπορία. Η Ευρωπαϊκή, Οργάνωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που πάει σε εμπορία κάθε χρόνο. Ε, το πληρώνει στην οργάνωση παραγωγών. Άρα αυτό είναι ελκυστικό. Θέλει κάποιος, θα θέλει να πάει κανείς σε μια τέτοια οργάνωση που προσελκύει η δημόσια χρηματοδότηση. Για τη σύσταση τώρα της οργάνωσης παραγωγών, αν δεν υπάρχει και θέλετε να τη συστήσετε, και γι' αυτό προβλέπετε χρηματοδότηση. Ε, αλλά όπως είπατε πολλοί από εσάς, όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Γιατί η προσφορά δεν γίνεται ευρύτερα δεκτή. Συμφωνώ εδώ με τον κύριο Ντόρφμαν σε μεγάλο βαθμό είναι ένα εθνικό θέμα, είναι, έχει ιστορικές ε, ε, εξηγήσει και δημιουργεί μια κουλτούρα που δύσκολα μπορούμε εμείς να την αλλάξουμε από τις Βρυξέλλες. Χρειάζεται χρόνος, είμαστε πεπισμένοι ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση σύν χρόνο, αλλά η διαδικασία είναι μακροπρόθεσμη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, εκτός από τη βοήθεια αυτή και τα κράτη-μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν επιπροσθέτως. Και αυτό το εξετάζομαι. Πρόσθετη ενίσχυση από τα κράτη-μέλη για να δώσουν κίνητρα στη δημιουργία των οργανώσεων παραγωγών. Μάλλον θα χρειαστεί κάτι περισσότερο όμως. Μια ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανταλλαγή πληροφοριών ούτως ώστε οι οργανώσεις των παραγωγών και η, παρα... εθνική παραγωγή που είναι καλά οργανωμένη να μιλήσουν σε παραγωγούς άλλων χωρών και να δημιουργήσουν ένα σύστημα αλληλοβοήθειας και βελτίωσης της υφισταμένης κατάστασης. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση θα είναι η απλούστευση. Ε, πολύ το είπατε. Απλοποίηση. Πρέπει να γίνει απλοποίηση. Ε, να γίνει απλούστερη διαδικασία σύστασης οργάνωσης παραγωγών. Αυτά κύριε Πρόεδρε είχα να σας πω στο τέλος αυτής της συζήτησης και βέβαια χαιρετίζω το γεγονός ότι έγινε η εκθεσή αυτή και θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω επ' αυτής μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα λόγος και πάλι στον ε, συνάδελφο κύριο Μέλο. Παρακαλώ χρόνο φίδου γιατί έχει ήδη καταφτάσει ο επίτροπο να μην τον αφήσουμε να περιμένει πολύ. Άλλωστε μην ξεχνάτε θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Θα είμαι λακωνικός γιατί όπως είπα η πρόθεσή μου ήταν να ακούσω περισσότερο τους συναδέλφους ε, και να συγκεντρώσω τις προτάσει και τι στάσεις του που θα είναι χρήσιμες για τη σύνταξη της έκθεσής μου. Το σημαντικό είναι ότι όλοι συμφωνούμε ως προς τη διάγνωση. Και όλοι έχουμε επίγνωση ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να βελτιωθεί η οργάνωση των παραγωγών προκειμένου να συσπυρώνονται και να οργανώνονται πολύ περισσότερο σε οργανώσεις. Γιατί είναι, όπως είπε ο κύριος Ντόρφμαν, η κατάσταση είναι ε, διαφορετική από χώρα σε χώρα και ίσως είναι και πολιτισμικό το θέμα. Η κάθε χώρα ε, έχει ξεκινήσει ανάλογα με τις ανάγκες της ε, το καθεστώς αυτό. Άλλες χώρες έχουν μακρόχρονη παράδοση οργάνωσης, άλλες χρειάστηκε να ξεκινήσουν εκ του μηδενός. Επίσης υπάρχει θέμα αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της κατάστασης. Σε ορισμένες χώρες δημιουργήθηκαν οργανώσεις παραγωγών, αλλά δεν ήταν βιώσιμες επειδή δεν κατάφεραν να διαχειριστούν καλά την κατάσταση. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να θεωρηθούν ελκυστικές οι οργανώσεις των παραγωγών από τους παραγωγούς. Κανένας παραγωγός δεν θα προσχωρήσει σε μία οργάνωση αν δεν δει ωφέλη από τη συμμετοχή σε αυτή αν δεν ε, δει προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή. Όποιο και είναι το μέγεθος του παραγωγού. Θα πρέπει να δει ωφέλη ε, στην οργάνωση για να προσχωρήσει αυτή. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς ε, μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, θα πρέπει να πούμε στους γεωργούς ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τη γεωργία, να οργανωθούν σε οργανώσεις παραγωγών και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. διαπιστώσαμε κάποιες αδυναμίες, κάναμε διάγνωση, εναπόκειται σε εμά να αντλήσουμε συμπεράσματα και να προτείνουμε μέτρα βελτίωσης. Θα πρέπει να δείξουμε τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού των οργανώσεων. Άλλοι έχουν μεγάλες εκμεταλλεύσεις, άλλες μικρές, αλλά οι συνθήκες ανταγωνισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί οι οργανώσει παραγωγών μπορεί να γίνουν σημαντικό μηχανισμός που θα ωφελήσει τους ε, Γιώργους, παρόλο που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα κάτι τέτοιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ισπανία, όπως ακούσαμε, έχουμε πολύ ικανές οργανώσεις παραγωγών και εξαιρετικά αποτελεσματικές. Και μιλούμε για τη Νότια Ευρώπη. Έχουμε παραδείγματα και προς μίμηση, αλλά και προς αποφύγη και στη Βόρεια Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε από όλα αυτά τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είχαμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση, δεν σας περιόρισα καν χρονικά, είχατε την ευκαιρία όλοι να λάβετε το λόγο. Είχαμε πραγματικά μια πολύ καλή συγκυρία και την πολυτέλεια χρόνου και ολοκληρώσαμε και εγκαίρως το θέμα αυτό. Είμαστε έτοιμοι τώρα να υποδεχθούμε τον Επίτροπο. Otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia. Ε, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Γεωργίας τον νέο μας Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Φιλ Χόγκαν. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε με τον Επίτροπο ήταν στην ακρόασή του της Δευτέρας Οκτωβρίου. Καλωσορίζω και τον Γενικό Διευθυντή και πολλούς από την Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θερμό καλωσόρισμα προς όλους. Θα ήθελα κύριε Επιτρόπη να σας πω ότι μετά την τελευταία μας συνάντηση και την ακρόαση όπου κρίναμε την επάρκεια των γνώσεών σας και τη συνάφεια του οράματός σας για την Γεωργία νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα των ιδεών μας και των δεσμεύσεών μας κατά την αντιμετώπιση των τρέχουσων και μελλοντικών προκλήσεων της Γεωργίας. Δεν θα ήθελα να προδικάσω τη συζήτηση, θα αφήσω τους συναδέλφους να θέσουν τις ερωτήσεις τους, που φαντάζομαι θα αφορούν διάφορες πτυχές του χαρτοφυλακίου σας. Θα μιλήσουμε για πολλά επίκαιρα θέματα, αλλά και για το όραμά σας για την γεωργική πολιτική. Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα ασχοληθούμε λοιπόν με πολλά και διάφορα θέματα. Χθε, για παράδειγμα ε, επισήμανα ε, στη συνάντηση που είχαμε με το Σώμα των Επιτρόπων στην διάσκεψη των ε, Προέδρων Επιτροπών ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θεωρώ ότι η γεωργία και ο γεωργικός κλάδος δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής στην παρουσίαση των 10 προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ θεωρώ η κοινή γεωργική πολιτική είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι λειτουργεί τόσο εύρυθμα ώστε δεν χρήζει πια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ δυσκολίε στην εφαρμογή τη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τη νέα κατάσταση και στην κοινή γεωργική πολιτική. Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή της ε, ΚΑΠ. Το θέμα της ε, δυσκολής εφαρμογής, ε, ιδιαίτερα για το πρασίνισμα. Χρειαζόμαστε περαιτέρω απλούστευση του καθεστώτος. Επίσης, θα πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα για να λάβουμε υπόψη της, την κρίση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της απαγόρευσης εισαγωγών της ρωσικής κυβέρνησης. Αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, αλλά έχουμε και τη διαφαινόμενη κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα και την κρίση στον απορροκυπευτικό τομέα στις χώρες Βαλτικής, στην Πολωνία, εξαιτίας του ρωσικού εμπάργου. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια νέα αγορά, άρα τα προβλήματα δεν είναι τοπικά ούτε εθνικά. Επίση, έχουμε τι προκλήσει που θα δημιουργηθούν από τι διαπραγματεύσει μα στην DTIP, τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορία και Επενδύσεων. Θα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα συμφέροντα των γεωργών και τη σημασία τη γεωργία και στι διαπραγματεύσει αυτέ. Επίση, ε, κύριε Επίτροπε, να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σα. Θα σταθούμε στο πλευρό σας και θα σας στηρίξουμε στο δύσκολο αυτό έργο σας και στις δύσκολες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε. Γιατί στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε από κοινού τα συμφέροντα της γεωργίας, την ασφάλεια των τροφίμων και την εύρυθμη εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής. Αυτά από μένα κύριε Επίτροπε. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, όπω σα είπα πριν από δύο μήνε, έχει αναλάβει δέσμευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα ε, συζήτησης ε, τη ε, πολιτική στο μέλλον. Η γεωργία, η, ανάπτυξη, η αγροτική ανάπτυξη είναι στο ε, επίκεντρο της πολιτικής της καινούργιας ε, Κομισιόν και με τον Επίτροπο Κατάινενε και με την ομάδα του συζητώ και συνεργάζομαι. Έτσι λοιπόν ο στρατηγικός τομέας η Γεωργία θα συμβάλλει ε, σημαντικά στη νέα, στο νέο οικονομικό θεματολόγιο. Ορισμένα βασικά στοιχεία είναι τα εξής. 25 εκατομμύρια είναι οι αγρότες, 50% είναι οι αγροτικές περιοχές. 7% παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα τροφίμων και 3,5% είναι η προσθέμενη αξία. Ε, οι αγροτικές περιοχές 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ε, της αυξηνόμενης ε, ζήτησης για τρόφιμα εμείς έχουμε αύξηση εξαγωγών τα προηγούμενα πέντε χρόνια που είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι οι εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων από την Ένωση. Ε, έτσι λοιπόν υπάρχουν ανάντι και κατάντι ε, συνδέσεις και με άλλου τομείς, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, λοιπάσματα για να μην μιλήσω και τον κεντρικό ρόλο που παίζει, οικονομική, ε, παίζει για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Η νέα ΚΑΠΑ δίνει μεγάλη ευκαιρία μεγιστοποίηση τη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ε, εξυγχρονισμός του τομέα με προσανατολισμό στην αγορά, νέες αναπτυξιακές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές, θα βοηθήσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και με την μεγαλύτερη έρευνα θα υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση για την αύξηση της παραγωγικότητας για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη δυναμική του γεωργικού τομέα σε ό,τι αφορά επενδύσεις, ανάπτυξη, απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την χρηματοδότηση για τους αγρότες, κυρίως τους νέους αγρότες, όπως ε, όταν αρχίζουν ε, στα διαδρομία τους και δουλεύουμε σε συνεργασία στενή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι σημαντικοί οι νέοι αγρότες για το μέλλον της ΚΑΠ, της ανταγωνιστικότητας, της ε, ανάπτυξης απασχόλησης. Ε, πολλές φορές ε, είναι γυράσκουσα, ε, γυράσκον ο πληθυσμός των γεωργών και είναι μετριοπαθής η βελτίωση. Ε, η ΚΑΠ έχει ιστορία πέντε ετών. Ο πρώτος πυλώνας ε, έχει ένα συγκεκριμένο μέσο για να στηρίξει τους νέους αγρότες ε, που είναι υποχρεωτικό δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη. 25% πρόσθετε σε ενισχύσεις για τα πρώτα πέντε έτη υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά μέτρα στήριξης για τους νέους στα πλαίσια της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στα πλαίσια επιχειρησιακού σχεδίου μέχρι 90% καλύπτονται οι επενδύσει. Ε, υποστήριξη για την εκπαίδευση, ε, κατάρτιση και συνεργασία. Η μεταφορά γνώσης λοιπόν στην πράξη μπορεί να επιδιωχθεί ε, μέσα από συμπράξεις για την καινοτομία, την παραγωγικότητα και με όλα αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η γεωργία ελκυστική απασχόληση. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διερευνήσουν τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που υπάρχουν στα πλαίσια πλαίσια των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ΠΑ, ούτως ώστε να υπάρξουν αυξήσεις στους ε, δικαιούχους. Στο Horizon 2020 και πρόσφατα είπα και για την ε, εταιρική σχέση για την καινοτομία θα ενθαρρύνουμε την ε, έρευνα και ανάπτυξη και πρόσβαση στη χρηματοδότηση των νέων. Αυτά είναι βασικά εργαλεία τα επόμενα χρόνια που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα βοηθήσουν μια γεωργία με βάση τη γνώση. Θέλουμε να μπορούμε να ε, έχουμε ε, περισσότερη απασχόληση σε ένα βιώσιμο περιβάλλον ε, για να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις προκλήσεις. Η απλοποίηση είναι η κορυφαία προτεραιότητα για το πρόγραμμά μου μέχρι το 2015. Η γραφειοκρατία μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στη λήψη αποφάσεων απλούστεροι κανόνες αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, τη δυναμική της γεωργίας και το εμπόριο στη γεωργία. Γι' αυτό πρέπει να απλοποιήσουμε τους ε, κανόνες, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία αποτελεσματικά, να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε ευέλικτοι στην προσέγγιση μας. Η απλοποίηση δεν μπορεί να γίνει μια ανοιχτή, ούτε θα γίνει κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι μια συνεχής ε, βελτίωση ε, οι μικρά και μεγάλα βήματα για να διευκολύνουμε τη ζωή των γεωργών. Πρέπει να τα κάνουμε αυτό όπου είναι δυνατόν και το ταχύτερο δυνατόν για να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο και να γίνει πιο προσοδοφόρος και ανταγωνιστικό στο τομέα της γεωργίας. Αυτό θα πρέπει να διέπεται από τις εξής αρχές κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, επειδή το επίκεντρο της περιοχής μας είναι οι αγροτικές περιοχές και οι αγρότες θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε τους ε, κανόνες προς το συμφέρον τους, ώστε να υπάρχει σταθερότητα ε, για τους δικαιούχους και τις εθνικές αρχές. Έτσι θα μειωθεί και το ο διοικητικός φόρτος. Η απλοποίηση για μας επικεντρώνεται στα στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν στα πλαίσια του παρόντος πλαισίου, πολιτικού πλαισίου. Η για να έχουμε καλύτερη Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Όλοι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με εθνικές και περιφερειακές αρχές, τους δικαιούχους και τους εμπλεκομένους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κρίνουν καλά την υλοποίηση επιτόπου των μέτρων της ΚΑΠ. Θέλουμε την πείρα τους, θέλουμε τις προτάσεις από τη δική του στην πλευρά για την απλοποίηση. Γι' αυτό το λόγο σας ενθαρρύνω αξιότιμα μέλη να αρχίσετε συζήτηση με την, στις εκλογικές σας περιφέρειες και να μας δώσετε βελτιωτικές ιδέες, συστάσεις. Είστε οι οι ε, κλεγμένοι αντιπρόσωποι των ε, Ευρωπαίων Γεωργών. Ε, συνεργαστείτε μαζί μου για αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη, οι ευρωβουλευτέ, οι γεωργοί, οι κομισιόν. Μπορούμε το 2015 να δώσουμε τα παραδοτέα που πρέπει. Πρώτη θέμα θα επίση, κύριε Πρόεδρε, να θέσουμε αυτό το σημαντικό θέμα στι 15 Δεκεμβρίου στα κράτη-μέλη, στα πλαίσια του Συμβουλίου. Ήδη ε, αρχικάναμε ε, μια διαδικασία ελέγχου της αγροτικής πολιτικής για να δούμε τι απλουστευσή μπορεί να γίνει και παράλληλα με την αρχή της επικουρικότητας. Και, δηλαδή εκεί τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι πρέπει να κάνει το κράτη-μέλη. Ε, τώρα αυτή τη διαδικασία ελέγχου την ε, έδωσε αποτελέσματα τα οποία αξιολογούμε. Βλέπω τέσσερις σημαντικούς τομείς όπου πρέπει να πλουστευτούν οι κανόνες τους επόμενους μήνες και έτη. Πρώτον, πρέπει να προ... κάθε πρόταση ε, θα πρέπει να ε, δίνει αποτελέσματα και στη νομοθετική διαδικασία θα πρέπει η απλοποίηση να ενισχύεται. Πάνω από 200 κανονισμούς που εφαρμόζουν την κοινή οργάνωση αγοράς θα αναθεωρηθούν. Αυτό το εγχείρημα είναι που θα πλουστεύσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις στον τομέα ε, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ε, τρίτον, ε, το νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων. Βεβαίως, ε, η προηγούμενη Επιτροπή ήθελε να, το να ξαναδεί τους κανόνες μετά το πρώτο έτος της εφαρμογής τους. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί, θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να απλοποιήσουμε τους άλλους κανόνες του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων για να μην ξαναρχίσουμε, να μην όμως την πολιτική συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις το, όπως έχουν επικυρωθεί από εσάς. Τέταρτον, θέλουμε να δούμε καλά τους κανόνες για γεωγραφικές ενδείξεις. Οι γεωγραφικές ενδείξεις βοηθούν τους παραγωγούς τροφίμων να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να αυξάνουν την απασχόληση επί τόπου. Θέλουμε να συνεχίσουν να αυξάνονται. Ε, θέλουμε αποτελεσματικούς κανόνες και όσο γίνεται απλούστερους. Ε, είμαι βέβαιος ότι όταν συνδυάσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες θα κάνουμε μεγάλη διαφορά τα βελτίο για τους αγρότες και θα μειώσουμε και το διοικητικό φόρτο για τα κράτη-μέλη. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα στην κατάσταση της αγοράς. Άκουσα τα ανησυχίε σας και ορισμένες προκλήσεις θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις λύσουμε. Καταρχήν γνωρίζω πολύ καλά ότι ε, στο γαλακτοκομικό τομέα ε, χειροτερεύει η κατάσταση στην αγορά και από την ρωσική απαγόρευση που επηρέασε τους παραγωγούς. Τώρα πρόσφατα η Κομισιόν πήρε και άλλα μέτρα για την αγορά που παρατείνουν την διαθεσιμότητα της ιδιωτικής αποθεματοποίησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2015 και αυτό είναι σημαντικό, ούτως ώστε να έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας που θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς. Επίσης ε, εγκρίναμε και στοχευμένη υποστήριξη για τους γαλακτοπαραγωγούς και θα παρακολουθούμε πολύ καλά τις αγορές που επηρεάζονται από τον αποκλεισμό. Επίσης ε, ε, η οικονομική κατάσταση παρακολουθείται ιδιαίτερα στα προϊόντα, όπως επηρεάζει τα προϊόντα ε, που επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργο. Ε, θέλουμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά παραγωγούς και αγρότες και θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει τεράστια γεωπολιτική και οικονομική σημασία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Όπως γνωρίζετε, τα σημερινά μέτρα συμπεριλαμβάνουν μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς ε, για τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα, τα οποία ε, οδήγησαν σε απόσυρση 93 τόνων από την αγορά. Θέλουμε να βρούμε νέες, προ... νέες αγορές για αυτά τα προϊόντα. Θέλουμε για τα ευαλείωτα να βρούμε αγορές ε, ε, από... για να ε, αντιμετωπίσουμε τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά. Άλλο ε, μέτρο στοχευμένο στις 29 Σεπτεμβρίου ε, θα λήξει το τέλος του 2014. Πάνω από 100.000 τόνοι προϊόντων αποσύρθηκαν με βάση αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, για να παρουσιάσω μια πιο αισιόδοξη θετική εικόνα. Όταν συγκρίνουμε το Σεπτέμβριο του 2014 με το Σεπτέμβριο του 2013, η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκε κατά περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό επιβεβαιώνει και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμόζεται στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα και να βρίσκει εναλλακτικού προορισμούς για τα προϊόντα της. Επίσης, η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση φαίνεται να είναι ε, ένα στοιχείο που προωθεί την γεωργία μας. Ε, εμείς θέλουμε να έχουμε καλή προστασία για υψηλής αξίας προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, ε, τώρα διαπραγματευόμαστε διμερώς πολλές συμφωνίες μαζί και την ε, TTIP, Διατλαντική Συμφωνία. Θέλουμε και άλλες αγορές να ανοίξουν στα υψηλής ποιότητας προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε όμως τα προϊόντα μας στο βωμό κάποια συμφωνίας. Τώρα γίνονται ε, ε, συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης η λειτουργία της ε, αλυσίδας των τροφίμων. Ε, έχουμε ε, προβλήματα με τη διαπραγματευτική δύναμη των γεωργών. Υπάρχουν ανισορροπίες δηλαδή στην δυνατότητα διαπραγμάτευσης των γεωργών. Αυτό θα το δούμε και θέλουμε να βελτιώσουμε την διανομή της προσθέμενης αξίας στην αλυσίδα των τροφίμων και εφοδιασμού. Ε, και θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο εδώ. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα την τελευταία φορά που ήρθα εδώ ότι θα εξετάσω κάθε εναλλακτική και προτάση νομοθετικού περιεχομένου για να αντιμετωπίσω προβλήματα στην αλυσίδα τροφίμων. Τώρα, σε προγράμματα ανάπτυξη, έχουμε πάρει 116 από 118 προγράμματα ήδη και περίπου 80 επιστολές ε, με παρατηρήσεις εστάλησαν στις διαχειριστικές αρχές. Φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο όπου σύντομα το πρώτο πρόγραμμα θα εγκριθεί. Οχτώ προγράμματα θα, θα, εγκριθούν μέχρι το τέλος του ε, έτους. Ε, ορισμένα δεν θα εγκριθούν αλλά θα είναι έτοιμα. Και θα γίνει η διαδικασία μεταφοράς ε, που θα ολοκληρωθεί το... πριν από το Μάρτιο του 2015. Τα άλλα προγράμματα θα γίνουν μετά την αναθεώρηση του MFF και στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η καθυστερημένη έγκριση του MFF και ο σχετικός κανονισμός επηρεάζουν πολύ την ικανότητα των κρατών μελών να υποβάλουν το 2014 προγράμματα. Οι περισσότεροι τα έδωσαν το δεύτερο εξάμεινο αυτού του έτους μέλη της Επιτροπής σας έκανα μια ανασκόπηση της, ε, του θεματολογίου απλοποίησης και τα μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς, ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και την πρόοδο διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τη σημασία του να δούμε τις αδυναμίες και να τις λύσουμε στην ε, αλυσίδα των τροφίμων. Με την υποστήριξή, μας, υποστήριξή σας θα συνεργαστούμε για να ε, δημιουργήσουμε ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ανταλλαγή απόψεων τώρα. Πρώτα θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Δυστυχώς έχουμε λίγο χρόνο. Δύο λεπτά λοιπόν οι συντονιστές σε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Κατόπιν θα απαντήσει ο Επίτροπος και στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων οι ομιλητέ θα δικαιούνται ένα λεπτό μόνο για τις παρεμβάσεις τους. Λυπούμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. που πήγατε και στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή μας απόψε, την πιο σημαντική ε, για τα θέματά σας. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε καλά. Έχω μια μεγάλη ανησυχία. Πολλοί αγρότες δεν ξέρουν ακόμα πώς θα εφαρμοστεί η αγροτική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και η Κομισιόν ακόμα γράφει ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ε, να μην γίνει νομότυπα δηλαδή σύνομα η μεταρρύθμιση. Λέει ότι, το, και παραθέτω, το γεγονός ότι... Ε, ε, ε, έλεγχη στις εκτάσεις των κρατών μελών ε, είναι δύσκολη, ότι είναι ψηλό το ποσοστό των ε, σφαλμάτων στο δεύτερο πυλώνα από το σύστημα ισοδυναμίας, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή η ίδια η Κομισιόν, η Γενική της Διεύθυνση, εκφράζει μεγάλες ανησυχίες ότι θα έχουμε ε, ε, δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος. Τι θα κάνετε εσείς κύριε Επίτροπε, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούμε τόσο πολύ στο μέλλον, τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε προβλήματα, ε, τη διόνυση των προβλημάτων σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Δώσατε πραγματικά εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου. Κύριος Δεκάστρο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Με χαρά μας σας βλέπουμε εδώ σήμερα υπό την επίσημη ιδιότητά σας. Όπως ξέρετε έχει μεγάλες προσδοκίες από το πρόσωπό σας ε, η Επιτροπή. Λοιπόν, ε, είναι καλό το πρόγραμμα για τους νέους, η πρόσβαση στις ενισχύσεις και εδώ θα βρείτε για όλα αυτά στην Επιτροπή μας ένα σίγουρο σίγουρο σύμμαχο στη μάχη σας κατά της γραφειοκρατίας και στη μάχη σας για την απλούστευση. Εδώ Έχουμε επικραθεί που μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που κάναμε στην προηγούμενη θητεία ε, έφερε περισσότερο γραφειοκρατικό βάρος και όχι λιγότερο και αυτό είναι μια ανησυχία ε, που μας δημιουργεί όσον αφορά και την εφαρμογή του πρασινίσματος που θέλουμε αλλά μας προβληματίζει όταν διαβάζουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι του 7-8% σφαλμάτων στην εφαρμογή του πρασινίσματος, του greening. Και αυτή είναι μεγάλη ανησυχία μας δημιουργείται. Θέλουμε ένα greening που εφαρμόζεται αλλά δεν θέλω να χάνουμε 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις. Μετά, κύριε Επίτροπε, η κατάσταση του γάλακτος είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πιστεύουμε ότι θα επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, θα επιδεινωθεί διότι η τάση λόγω της δραματικής μεταβολής των τιμών οδηγεί σε πολύ μεγάλες κρίσεις σε πάρα πολλές ε, χώρες της Ευρώπης. Ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε ε, τι γίνεται σε, αυτό το, σε αυτή την μετάβλητη κατάσταση μετά τις ποσοστώσεις. Το συζητήσαμε πολύ και δεν κάναμε σχεδόν τίποτα. Θέλουμε καινοτομίες, θέλουμε ιδέες, ε, νέα μέσα για τη διαχείριση του κινδύνου και για να διαχειριστούμε αυτό τον μετάβλητο χαρακτήρα των τιμών ο τομέας ε, των, ε, της τυροκομείας ε, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όμως υπάρχουν και θετικά νούμερα που τα παραθέσατε. Για μία ακόμη φορά σας το λέω, χρησιμοποιήστε αυτή την Επιτροπή σαν ισχυρό όμα, όπλο για να ενισχύσετε τους ε, δεν υπάρχει αντιπαράθεση, έχουμε βούληση να δράσουμε, να κάνουμε κάτι και ελπίζουμε αυτή η δράση να, λάβει η χώρα το ταχύτερο δυνατόν, να κινητοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Σνίκολσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ με τις απόψεις που ακούστηκαν για το πρασίνισμα. Ε, το θέμα είναι ότι το λεκτικό συνέδριο θα είναι υπεύθυνο για το πρασίνισμα και το λεκτικό συνέδριο δεν έχει όλε τι γνώσει όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Σα παρακαλώ αυτό να το έχετε υπόψη. Δεν θέλουμε αυτό το πρόβλημα να επιληθεί το 2016 ή το 2017. Θέλουμε να λυθεί το 2015. Λοιπόν, να αναφερθώ σε αυτό που θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία στην ε, Ευρώπη. Είναι η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα ε, συνέβη, ξέρουμε το ιστορικό, το υπόβαθρο γιατί συνέβη. Κύριε Επίτροπε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και έχετε κι εσείς, είναι η δυνατότητα να αναθεωρήσουμε και να αυξήσουμε την ε, τιμή παρέμβασης. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που έχετε στη διάθεσή σας. Ε, δεν είναι ρεαλιστικό το επίπεδο το τωρινό και είναι ένα άχρηστο εργαλείο στην εργαλειοθήκη που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Αναθεώρηση λοιπόν της παρέμβασης, της τιμής παρέμβασης θα βοηθούσε τελικά ε, να ανακάμψει η αγορά. Και στην προηγούμενη ε, κρίση του 2008 και του 2009 είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ποτέ ξανά δεν θα επιτραπεί να διαρκέσει τόσο πολύ μια κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Παρακαλώ μην πέστε στην παγίδα ε, προηγούμενων Ευρωπαϊκών Επιτροπών πιστεύοντας ότι όλα θα λυθούν την επόμενη άνοιξη. Κάποιοι μας λένε ότι θα μπορούσε να είναι το φθινόπωρο του χρόνου. Εγώ να σας πω τώρα ότι θα είναι εκτός δουλειάς η γεωργία του γαλακτοκομικού τομέα πριν το επόμενο φθινόπωρο. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα σύντομα. Καλωσορίζω αυτό που είπατε για τη συνεργασία με τις τράπεζες, διότι οι τράπεζες έχουν το ρόλο να παίξουν σε όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν τους γεωργούς να κινούνται μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι οι μεγάλοι ηλιανοπολιτές. Ε, είναι μόνοι τους τελικά όσον αφορά το πρόβλημα που δημιουργείται με την ε, μεταβολή των τιμών. Ευχαριστώ κύριε Ρόντε. Thank you, Mr. Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ και στη γραπτή απάντηση που δώσατε στην επιστολή που στείλαμε με τον κύριο Ντές Νίκολσον και Δεκάστρο για την αναβολή του greening της ΚΑΠ. Κατά κάποιο τρόπο αυτή ήταν η απάντηση που περίμενα από εσά. Γιατί φυσικά δεσμεύεστε από προηγούμενε αποφάσει. Αλλά επιτρέψτε μου ένα προσωπικό σχόλιο. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι, ως, ο, ότι εσείς ως νέος επίτροπος μα, γύρατε πολλές ελπίδες και προσδοκίες και μετά την τελευταία μας ακρόση έλεγα αριστερά και δεξιά πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε ως νέο Επίτροπο Γεωργία τον κύριο Χόγκαν. Γιατί, Γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε αλλαγή στην προσέγγιση της γεωργίας και του γεωργικού κλάδου στην Ευρώπη. Γι' αυτό και απογοητεύτηκα με την απάντηση που μας στείλατε. Γιατί είναι η απάντηση του συστήματος, όχι η απάντηση του πολιτικού, όχι η απάντηση του κυρίου Χόγκαν του Επιτρόπου, ούτε μια απάντηση για τους γεωργούς. Ε, το σύστημα παντά ας μείνουμε στα συμπεφωνηθέντα και σε ανηλυμένες υποχρεώσεις και σε αυτό που προβλέπει το σενάριο. Θα δημιουργήσετε όμως ένα γραφειοκρατικό τέρας στο πρασίνισμα της γεωργίας και θα ε, ενισχυθεί η άνηση εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όλοι το βλέπουν αυτό. Είναι πασιφανές. Ερωτώ λοιπόν, αν δεν θέλετε να αναβάλλετε το πρασίνισμα της ΚΑΠ, πείτε μας τουλάχιστον πώς θα αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία και την ανομοιόμορφη ή άνηση εφαρμογή αυτού του τμήματος της ΚΑΠ. Και αυτό για χάρη των γεωργών. Θέλουμε να μας δώσετε κατάλληλες ε, και εύστοχες απαντήσεις για το θέμα αυτό. Αν όχι σήμερα, τουλάχιστον όσον ε, Ευχαριστώ. Η κυρία Σένρα. Ε, Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση μόνο. Κύριε Επίτροπε, είστε έτοιμος και πρόθυμος να αναθεωρήσετε τις πολιτικές και να θεσπίσετε κάποια μέτρα για τη ρύθμιση της παραγωγής και τη ρύθμιση των αγορών. Είναι σαφές ότι το πρόβλημα του γάλακτος δεν οφείλεται μόνο στο ρωσικό εμπάργο, στη ρωσική επαγόρευση, το πρόβλημα στο γαλακτοκομικό τομέα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην λήξη των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που προκάλεσαν μια σημαντική αύξηση της γαλακτοκομικής παραγωγής. Ευχαριστώ. Äh, Κύριε Επίτροπε, ε, μας είπατε πολλά πράγματα, αλλά δεν άκουσα για συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή ε, η απλοποίηση δεν αυξάνει ε, τα έσοδα των ε, γεωργών, ούτε αποτελεί αλλαγή της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα τι θα κάνετε. Γιατί φοβάμαι και οι συνάδελφοι των μεγάλων ομάδων που υποστήριξαν την μεταρρύθμιση ότι με την απλοποίηση ε, ε, ε, υπάρχει περίπτωση με την, το, πρασίνισμα να καταργηθεί μέσα από τη μεταρρύθμιση και την απλοποίηση. όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Για το γάλα, θα περίμενα μια απάντηση σήμερα. Ψάχνετε νέες αγορές για να πάνε τα πλεονάσματα εκεί. Πού θα βρεθούν ξαφνικά. Δηλαδή όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες γάλακτος πού θα πάνε με την πολιτική που δεν την αρχίσατε εσείς της απελευθέρωσης ε, του τομέα ε, με τις ε, εξαγωγικές ενισχύσεις, τις αποθεματοποίησεις, οδηγηθήκαμε σε ένα καθεστώς που πλήττει τον παραγωγό. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην αγορά ως λύση. Το TTIP προβάλλεται ως λύση για τις εξαγωγικές αγορές. Τις μελέτες που έχουν γίνει για τους κινδύνους τις ξέρετε, που τους έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα για τους ε, αγρότες στον τομέα του κρέατος. Δεν είναι στρατηγική, δεν είναι πανάκια δηλαδή τα TTIP. Δεν θα ωφεληθεί ολόκληρη η γεωργία στην Ευρώπη. Αντίθετα, επίσης θα περίμενα να πείτε συγκεκριμένα κάποια μέτρα μεσούσης της κρίσης. Η κρίση δεν επίκειται, είναι εδώ. Οι τιμές γάλακτος ε, πάνε προς την κατεύθυνση των 20 cents, άρα χρειαζόμαστε μια απάντηση. Όχι πρώτα θα κάνουμε την απλοποίηση και μετά τι θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι απάντηση αυτή, δεν συμβάλλει στην επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάγκνιου. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που θέλετε να πετύχετε απλούστευση. Θα σας ελέγξουμε αν το πετύχατε σε ένα χρόνο περίπου. Άλλο θεματάκι. Και θα δούμε πόσο πιστός είστε στις υποχρεώσεις που αναλάβατε. Οι Βρετανοί, οι Γεωργοί ανησυχούν γιατί μπαίνει πολύ Ιρλανδικό γάλα στην Βρετανία και ο πελάτης δεν μπορεί να κάνει διάκριση. Ποιο είναι Βρετανικό και ποιο είναι Ιρλανδικό. Αλλά είστε επίτροπος, πρέπει να ξεχάσετε τη χώρα από την οποία προέρχεστε. Για τους κανόνες για βιολογική καλλιέργεια στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειαζόμαστε αλλαγή. Είναι ένας τομέας ε, που μεγάλωσε, έχει μια μικρή αγορά, 4% περίπου, υπάρχουν κανόνες, συμμορφώνονται οι βιολογικοί γεωργοί και όλοι πρέπει να ζήσουμε κάτω από τον ίδιο ουρανό και δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος όσον αφορά τις προτάσεις. Η αλυσίδα, ο κώδικας για τον εφοδιασμό των παντοπολίων και με τους δείκτες λειτουργεί αρκετά καλά αλλά δεν θέλουμε παρεμβάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε ικανοποιημένοι αν ακολουθήσουν ε, την θέση που ακολουθήσαμε εμείς άλλες χώρες. Στον αρρώσιμο τομέα χάσαμε τα συστατικά, τα ενεργά στα ε, Χάσαμε 430 30 συστατικά τελευταία 13 χρόνια. Εάν δεν μπορούμε να έχουμε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, πρέπει να χρησιμοποιούμε την εναλλακτική που είναι τα παρασιτοκτόνα. Και αν και αυτά μας τα πάρουν, άρα θα είμαστε βιολογικοί γεωργοί και δεν θα έχουμε αρκετό φαΐ. Την τελευταία φορά που σας μίλησα, να έχω και άλλο χρόνο πρόεδρε, διότι με διακόπτουν οι πράσινοι. Επίτροπε, επιτροπή, ησυχία παρακαλώ. Ε, Επίτροπε να επαναλάβω την πρόσκλησή μου ε, να έρχεται στις ανατολικές κομιτείες της ε, Αγγλίας να δείτε σοβαρή αρρώσιμη γεωργία και να δείτε τι προβλήματα έχουμε με τα μέτρα. Και όλο και περισσότερα να ψεκάζονται. Αυτό θέλετε, πράσινοι. Ε, και επίσης, μήπω να έρθετε στο εργοστάσιο στο δηληστήριο του State and Light της Ζάχαρης στον Τάμεση, διότι η νομοθεσία σας σας ε, καταστρέφει 850 θέσεις εργασίας και ευχαριστώ το κόμμα των Πρασίνων για τις διακοπές στην ομιλία μου. Δώστε pan te dodatkowe sekundy. Ε, αρκετό συμπληρωματικό χρόνο σας χορήγησα. Ολοκληρώσαμε το γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο με τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ. Καταρχήν, αγγίξατε μια ευαίσθητη χόρδη σε ό,τι αφορά το, τα κοντήλα της Γεωργίας και χαίρομαι που ασχολείστε με θέματα που θα συζητήσω με την Γενική Διεύθυνση, με, τη, με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και χαίρομαι για τη γνωμοδότηση και της, την πίεση που ασκείται. Και ξέρω ποιες είναι οι ανησυχίες σας για το greening, για το πρασίνισμα. Αλλά κύριε Ρόντε αυτές τις αποφάσεις τις, αποφ... εφαρμόσατε, το αποδείξατε. Ε, δεν μπορείτε να περιμένετε από μένα να αναβάλω κάτι που δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η του 2015. Θα πρέπει να δούμε αν λειτουργεί. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά όμως το πρασίνισμα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνα τις πολιτικές και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που σας απασχολεί τόσο πολύ. Οπότε κύριε Δες, κύριε Δεκάστρο, κύριε Ρόντε και κύριε Νίκολσον, εσείς μιλήσατε κυρίω για τον για το πρασίνισμα. Ξέρετε, της, δεν μπορείτε να ξέρετε ότι είναι ανομοιόμορφη η εφαρμογή του, γιατί δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή το πράσινισμα. Θα πρέπει απλώς να φροντίσουμε οι πολιτικές που εφαρμόζουμε να είναι λογικές, να χαρακτηρίζονται από κοινή λογική και τα κράτη-μέλη που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εφαρμογή των πολιτικών θα πρέπει να το κάνουν έχοντας επίγνωση των κατευθυντήριων γραμμών και των στοιχείων των πολιτικών. Νομίζω ότι ήμουν σαφής για το θέμα αυτό. Τώρα, για τις ε, περιοχές οικολογικής εστίασης. Θα τις αναθεωρήσουμε μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η εμπειρία των δικαιούχων, των κρατών μελών και των ευρωβουλευτών από την εφαρμογή των περιοχών ε, η οικολογική εστίαση. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ή να αναβάλω μια πολιτική που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, παραλαμβάνω. Κύριε Δεκάστρο, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Ιταλική Προεδρία που έθεσε ως ύψη προτεραιότητα το θέμα των νέων αγροτών. Και το προέταξε και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη Συμφωνία για την ΚΑΠ. Είναι σημαντικό να έχουμε νέο αίμα, νέους καταρτισμένους αγρότες που θα εμπλουτίσουν το γεωργικό κλάδο. Και τώρα για πρώτη φορά έχουμε κάτι τέτοιο στην κοινή γεωρική πολιτική, μέτρα δηλαδή υπέρ των νέων αγροτών. Βέβαια κύριε Ντές και Δεκάστρο κάνατε μια έκκληση για τις κυρώσεις. Δεν θα υποβληθούν πρόστιμα οι κυρώσεις για το πρασίνισμα της κοινή γεωρικής πολιτικής στην πρώτη διετία εφαρμογή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η πολιτική. Απλώς την πρώτη διετία δεν θα επιβληθούν πρόστιμα οι ποινέ. Οπότε ήταν σημαντική αυτή η υποχώρηση που κάναμε. Είναι σημαντικό. Ισχύει αυτή η υποχώρηση και δεν θα εφαρμοστούν κυρώσει και πρόστιμα κατά την πρώτη διετία. Το γάλα, σημαντικό θέμα. Η ρευστότητα των τιμών, η αστάθεια των τιμών ε, είναι όντω ε, δύσκολο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι η αύξηση του 5% της γαλακτοκομικής παραγωγής θα αλλάξει αισθητά την κατάσταση το 2014. Και αυτό είναι το επίπεδο αύξησης ε, ε, της παραγωγής που... αλλά και για το γάλα ισχύουν οι κανόνες και οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Μην μου θυμίσετε τι συνέβη το 2009. Δεν, δεν έχουμε σήμερα δυσκολίες παρόμοιες με το 2009, αλλά αντλούμε συμπεράσματα από εκείνη την εμπειρία και βλέπουμε τι μηχανισμούς έχουμε στη διάθεσή μας, τι εργαλεία και τι επιπλέον μέτρα μπορούμε να λάβουμε και μάλιστα γρηγορότερα χάρη στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Οπότε Γνωρίζω τις ε, ανησυχίες σας για το γάλα. Θα επαγρυπνώ και θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση. Και είμαι έτοιμος να αξιοποιήσω τους μηχανισμούς που έχουμε και την κοινή οργάνωση αγοράς για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα. Πάντως θα πρέπει και οι Γεωργοί να καταλάβουν ότι υπάρχουν κανόνες που συμφωνήσαμε από το 2008 για την κατάργηση της σταδιακή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες, γιατί είναι άδικο από αυτούς που τηρούν τους κανόνες ε, να ε, τιμωρούνται ενώ να επιβραβεύονται εκείνοι που αδιαφορούν για τους κανόνες. Οι περισσότερες χώρες ε, τηρούν τους κανόνες. Ελάχιστες τους παραβιάζουν. Και Μπορεί να έχουμε και ένα σημαντικό, μια σημαντική υπερπροσφορά, μην σας εκπλήσει κάτι τέτοιο χρειαστεί. Τώρα, η παρέμβαση είναι ένα από τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα δούμε τι μηχανισμού και τι μέτρα έχουμε στη διάθεσή μα και τι είναι κατάλληλο για κάθε περίπτωση. Και φυσικά στους δύσκολους αυτούς καιρούς είναι σημαντικό να εμπλέξουμε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και καλό θα ήταν να έχουμε συνεργασία τραπεζών και γεωργών για να μπορούν να παραμείνουν ε, στην αγορά η παραγωγή. Αναφέρθηκε από την κυρία Σέρνα το θέμα των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση μετά την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που στην αρχή θα, προκαλέσουν κάποια στάθεια τιμών, αλλά έχουμε τα μέσα ε, ρυθμίσης της αγοράς, θα τα χρησιμοποιήσουμε όπου δει. Κύριε Χόισλινγκ μου είπατε να καταθέσω προτάσεις εγώ για απλούστευση όταν ζήτησα από εσά να με βοηθήσετε για να καταλήξουμε σε μια δέσμη μέτρων για την απλοποίηση. Γιατί αν ε, σας έθετα προτελεσμένο γεγονότο σίγουρα θα μου ζητούσετε κάτι άλλο. Έχετε την ευκαιρία πάντως ε, να εμπλακείτε σε αυτή την προσπάθεια, να συνεργαστούμε και από την εμπειρία που έχετε από τη Γερμανία, από την ε, εκλογική σας περιφέρεια θα συμβάλλετε στις νέες προτάσεις έχουμε μία ξεχωριστή μονάδα πια στην ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ακριβώς για να συγκεντρώσουμε εμπειρία από τα προβλήματα. Δεν αποκλείω κανέναν από τη συζήτηση για το πώς θα επιφέρουμε αλλαγές, γιατί όλες οι εμπειρίες ε, και όλες οι γνώσεις μας είναι χρήσιμες. Σας προσκαλώ λοιπόν από κοινού να εργαστούμε γι' αυτό. Και για το 2015 η απλούστευση είναι προτεραιότητα. Θα είναι το έτος της απλούστευσης. Θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια δέσμη μέτρων για να απλουστεύσουμε τα πράγματα για τους γεωργούς, φυσικά τηρώντας τους αρχούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Κύριε Άγνιου, με εντυπωσιάζεται που, θε... που θέλετε ευρωπαϊκή σήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Εσείς δεν θέλετε καμία επέμβαση από, την... από τις Βρυξέλλες σε τέτοια θέματα. Ίσως μετά από την νέα κατάσταση έχουμε αντίστροφη ροή του γάλακτος. Στο τέλος θα γίνεται και εσύ πέραμαχος κυλής γεωργικής πολιτικής αν υποβάλλετε τέτοιες απαιτήσει. Σε ό,τι αφορά τη βιολογική γεωργία, γίνονται εκτενείς συζητήσει για τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα. Είμαι ότι είμαι πρόθυμο να συνεργαστώ με τον κύριο Χόισλινγκ, τον εισηγητή, αλλά και του και εισηγητέ για να προωθήσουμε την πρόταση για τη βιολογική γεωργία. Και Φυσικά δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε το σημαντικό έργο και την προεργασία που έχει γίνει. Δεν θα πρέπει να τα πετάξουμε αυτά στα σκουπίδια, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη γνώση που έχουμε ήδη συσσωρεύσει. Ήδη έχω ξεκινήσει συζητήσεις με κάποιες χώρες που έχουν προβλήματα και ανησυχίε. Θα πάω την επόμενη εβδομάδα και στι κάτω χώρες για να εμβαθύνω στο θέμα αυτό. Και αντί να πετάξουμε στα σκουπίδια μία πρόταση στην οποία συμμετείχατε κι εσείς για να καταρτιστεί, καλό θα ήταν να την αξιοποιήσουμε και να τη βελτιώσουμε. Θα είμαι ελαστικός, διαλλακτικός και με τη βοήθεια του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών που είναι υπέρ της πρότασης θα τη βελτιώσουμε. Γνωρίζω πάντως ε, τις ανησυχίες κάποιων κρατών μελών και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόοδο. Και θα πρέπει να δείξουμε καλή βούληση για τα βιολογικά προϊόντα και αν απλουστεύσουμε τη γραφειοκρατία, αν εναρμονίσουμε τους κανόνες, θα ωφελήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στην βιολογική παραγωγή. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα του κλάδου και σε καμία περίπτωση να μην επιδεινώσουμε την κατάσταση της βιολογικής γεωργίας. Επίσης, θα πρέπει να εγκριθεί το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, τις επόμενες 15 μέρες και ευελπιστώ ότι η βιολογική γεωργία θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το 2015. Για την ε, ζάχαρη και το σχετικό εργοστάσιο που είπατε, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στις μεταρρυθμίσεις για τον τομέα της ζάχαρης είναι πιο ειδικό το θέμα. Θα ασχοληθούμε με αυτό κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Σε ό,τι αφορά τα συστατικά των φαρμάκων και το, τις αρρώσιμες καλλιέργειες, πολύ ευχαρίστω να επισκεφτώ και εσάς. Πριν τα Χριστούγεννα θα πάω στις κάτω χώρες. Δεν έχω οριστικοποιήσει ακόμη όμως τον κατάλογο με όλες μου τις επισκέψεις. Είμαι πάντως ανοιχτός. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε 30 εγγεγραμμένους ομιλητές. Ένα λεπτό καθένας. Παρακαλώ δείξτε αυρότητα για να απομείνει κάποιος χρόνος και στον Επίτροπο για να απαντήσει. Η κυρία Εράνς Γκαρσία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για να μην επαναλάβω ερωτήσει που έγιναν ήδη, εγώ θα σας μιλήσω για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Επίτροπε γνωρίζετε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να προστατεύσουμε τον τομέα του μοσχαρίσιου κρέατος και το κρέατος πουλερικών στις διαπραγματεύσεις του TTIP. Επίσης, χρειαζόμαστε κανόνες ποιότητας και για τις ονομασίες προέλευσης. Υπάρχει στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου να χρησιμοποιούμε κάποια μέτρα για να αποφύγουμε σφετερισμό αυτών των μέτρων προέλευσης ε, γιατί σημαντικά ονόματα όπως Ριόχα, Χερές, Μάλαγα, Βίνο Δερεσέρβα. Είναι σημαντικοί αυτοί οι όροι και χαρακτηριστικές ποιότητες και ονομασίες προέλευσης. Το θέμα της υγιεινής διατροφής. Η Ισπανία ζήτησε να διευρυνθεί το σύστημα διανομής στα σχολεία των απορροκυπευτικών και του γάλακτος και να συμπεριληφθούν και το το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, γιατί για την ε, καρδιά είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι κύριε Επίτροπε που ήσταν άμεσά μας ε, σήμερα. Καταλάβατε τις ανησυχίες και τη φροντίδα μας που κατάλαβα την απαντήσεις που δώσατε. Φοβάμαι δυστυχώς ότι οι απαντήσεις που δώσατε δεν είναι στο ύψος του διακυβεύματος. Παρόλο που συμφωνούμε όσον αφορά ε, τη διάγνωση. Δεν είναι στο ύψος ε, να ανταποκριθεί στην κρίση του γάλακτος. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει προτάσεις όσον αφορά τη συζήτηση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Προτάσεις που απερίφθησαν τον, στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου. Χαίρομαι που οι προτάσεις αυτές θα μπορέσουν να αναθεωρηθούν. Πίσω από το γάλα βέβαια υπάρχει και το θέμα της κρίσης της αγοράς του βοήου κρέατος που θα ακολουθήσει την κρίση του γάλακτος. Αυτό βραχυπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα. Πρέπει ε, να, να δούμε τι γίνεται στη Βραζιλία και στη ΣΥΠΑ σήμερα. Εκεί τα πάντα κινούνται και αλλάζουν. Η απελευθέρωση των τελευταίων ετών μείωσε το μηχανισμό για τη διαχείριση αγοράς και έχουν γίνει ευμετάβλητες οι τιμέ. Το αναφέρατε. Άρα το μοντέλο της γεωργίας που θέλουμε για την Ευρώπη ποιο είναι. Θέλουμε να συντηρηθεί η απασχόληση και η γεωργία σε εύθραυστο περιβάλλον. Και ποιο είναι το μοντέλο το γεωργικό που θέλουμε. Το χρονοδιάγραμμα προβληματισμού για τις μεταρρυθμίσεις είναι κάτι επίκαιρο. Θα πρέπει να μας δώσετε στοιχεία ούτω ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια μελλοντική μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Ο κύριος Κούσμουκ, αν μπορείτε να τα καταφέρετε καλύτερα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Δύο ερωτήσεις όσον αφορά τα τρέχοντα θέματα. Πρόσον αφορά το ρωσικό εμπάργο, όλοι οι γεωργοί υποφέρουν και όχι μόνο οι γεωργοί που έκαναν εξαγωγές στη Ρωσία. Είχαμε μια κατάρρευση στα διά, στις τιμές των γεωργικών αγαθών ε, στην Πολωνία από 30 μέχρι 70% έχουμε μειώσει των τιμών και οι αποζημιώσεις πηγαίνουν σε εκείνους που καταστρέφουν ε, τα προϊόντα ή τα παραδίδουν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο σύστημα για αποζημιώσεις του χρόνου. Δεύτερον, έχουμε ένα μετριοπαθές πακέτο για το γάλα από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τα τρία βαλτικά κράτη και τη Φιλανδία για τέσσερις χώρες συνολικά. Η Πολωνία έχει υποφέρει εξίσου από το ρωσικό εμπάργκο Κατά μέσο όρο η μείωση των τιμών του γάλακτος ήταν της τάξης του 20%. Αλλά η Πολωνία δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο. Γιατί αυτό. Κύριε Πόλσον, επόμενη. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Κύριε Επίτροπε, Αναφερθήκατε πολύ σε καινοτομία, απλούστευση, ανάπτυξη και τον Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με θέμα την μεταποίηση των ε, φυτών στην ε, Ευρώπη. Μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό. Είναι κάτι σημαντικό και ίσως θα μπορούσε να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις οργανώσεις των γεωργών αλλά και με τους διάφορους εμπλεκόμενους του φορέα, αλλά και με διάφορους εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη, ε, διότι όλοι θέλουμε να καταβάλουν προσπάθειες. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Κύριε Δαντέν, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ κύριε, Προ... κύριε Επίτροπε. Να εκφράσω ένα συνέστημα. Όταν είμαστε στις εκλογικές μας περιφέρειες ε, δεν μπορούμε σε αυτά που μας παρουσιάζει μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις απαντήσεις που δίνει στις αρχές που χειρίζονται τα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα και τις αρχές που διαχειρίζονται τον πρώτο πυλώνα, δεν βλέπουμε την πολιτική που ψηφίσαμε εδώ. Έχω το συνέστημα ότι η διεύθυνση η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, πραγματικά χρειάζεται όλο το βάρος σας στο σώμα των επιτρόπων, ούτως ώστε να υπάρξει εκ νέου μεγαλύτερη δύναμη για έναντι των άλλων γενικών διευθύνσεων που τελικά τσιμπολογούν και παίρνουν από την ε, γεωργική πολιτική. Ο Κούκος έχει τη μανία να φτιάχνει τη φωλιά του στη φωλιά των άλλων. Λίγο πολύ αυτό αισθάνομαι ότι γίνεται με κάποιες γενικές διευθύνσεις και θα ήθελα ειλικρινά η Γενική Διεύθυνση της Γεωργίας να στηριχθεί ούτως ώστε η πολιτική που ψηφίσαμε τελικά είναι εκείνη που θα εφαρμόζεται επί και όχι μια άλλη πολιτική. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντότζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπατε. Κυρίως αφορούσαν το μέλλον, κάνατε τη διασύνδεση μεταξύ γεωργίας, θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Η γεωργοί του γαλακτοκομικού τομέα στην Βόρεια Ελλανδία θα απογοητευτούμε αυτά που είπατε. Παραδεχτήκατε ότι έχει δυσκολίε ο γαλακτοκομικό τομέα, αλλά είπατε τα προβλήματα που αντιμετωπίσετε. Στη Βόρεια Ιρλανδία ήδη η παραγωγή του γάλακτο παράγουν σε πολύ χαμηλέ τιμέ. Το μισό γάλα που λέτε σήμερα. Ε, ε, έπεσαν ακόμα περισσότερο τιμές στο παγκόσμιο εμπόριο του Γάλακτο. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντω παρέμβαση για το γάλα. Είναι πρόσδεκτο το ότι έχουμε ευρύτερο χρονικό περιθώριο μπροστά μας, αλλά οι τιμές του γάλακτος δεν σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Όσον αφορά τις αλλαγές των τιμών, αυτή ε, η διακύμαση των τιμών και το τρίτο τρίμηνο θα διαρκέσει του χρόνου και θα επιδεινωθεί λόγω της λήξης των ποσοστώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είσαστε ανοιχτοί τουλάχιστον να εξετάσετε την ιδέα μιας σταδιακής προσέγγισης στην ε, φιλελευθερωποίηση της αγοράς του τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπράνεν. Ένα λεπτό, μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ. Είναι γνωστό. Ότι η γεωργία επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος. Ισχύει επίσης ότι η γεωργία ε, είναι υπεύθυνη για πάνω από το 9% των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα σχετικά λίγα έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές αυτές. Το πακέτο για την ενέργεια το κλίμα περιέχει ένα εργαλείο, δηλαδή την απόφαση για την κατανομή της προσπάθειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εκπομπές αυτές, όμως τα κράτη-μέλη θέτουν προτεραιότητες άλλους τομείς ε, και κάνουν σχεδόν τίποτα για τη γεωργία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη θα εξασφαλίσει ότι οι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία τη Ευρωπαϊκή Ενώση θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επόμενα χρόνια και ότι τα κράτη-μέλη θα μειώσουν τι εκπομπέ αυτέ στα πλαίσια του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά τη δασική κάλυψη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ούτω ώστε να συλλαμβάνεται περισσότερο άνθρακα και έτσι τελικά οι αλλαγές χρήσεως της γης στον θεσοκομικό τομέα να γίνεται καλύτερα τόσο ώστε να μειωθούν τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος. Επίτροπε, συγχαρητήρια για την ανάλυση των καθηκόντων σας. Ελπίζω να μην σας λείπει ο πολιτικός κόσμος της Ιρλανδίας πολύ. Αν σας παρηγορεί, δεν λησμονηθήκατε, δεν σας ξέχασα. Έγινε μια μάζοξη 10 Δεκεμβρίου, γίνεται μια μάζοξη 10 Δεκεμβρίου στο Δευλίνο για να μιλήσουμε για σας, για την κληρονομιά που αφήσατε. Ένα ερώτημα που ίσως θα τα ακούσετε συχνά είναι για τις επιτόπιους, για τις επιτόπιους ενέχους στα αγροκτήματα. Προφανώς γνωρίζετε ότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίζετε το ότι είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές, να ξέρουν ότι φαγητό παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιοδήποτε τρόφιμο πληρεί τις ύψεις προδιαγραφές ποιότητας και βέβαια χρειάζονται κανονισμοί, γι' αυτό χρειάζονται έλεγχοι, ούτω ώστε αυτό να γίνεται. Πολλοί όμως γεωργοί μας λένε καθημερινά και εβδομαδία ότι οι παρούσες διαδικασίες είναι υπερβολικέ, ότι το Υπουργείο Γεωργίας το θεωρούν ότι είναι εχθρό του, ότι πάνε εκεί για να τους πιάσουν στα πράσα επιθεωρητές. Έχετε κάποια σχέδια, θα ξεκινήσετε κάποια διαβούλευση, ούτω ώστε η διαδικασία ελέγχων να γίνει πιο διαφανής και πιο δίκαιη στα μάτια και των γεωργών αλλά και των καταναλωτών. Ε, κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τα σχόλια που κάνατε για αυτό το νόμο, για το μεγάλο φόρο. Είπατε ότι είναι τρελό ότι πρέπει να πληρώσουν τεράστιους λογαριασμούς, ε, δύσκολους καιρούς κάποιες αγορές, κάποια γεωργοί. Μήπως ε, μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Ίσως είναι εθνικό το θέμα. Τα ερωτήματα όμως που δημιουργεί τη σχέδια αναπτύξεως υπαίθρων προβληματίζουν. Λοιπόν, για το Ιλλανδικό σχέδιο αναφέρονται η κοινή προσέγγιση ότι 50% συμμετοχή ελάχιστη πρέπει να υπάρχει. Φαίνεται δεν απαραίτητο, μπορείτε το διευκρινίσετε, διότι πολλοί γεωργοί στη γεωργία στους διάφορες ορεινές περιοχές προβληματίζονται. Τώρα για τι ανησυχίε των Βρετανών ε, γεωργών έναντι των Ιρλανδών. Εμείς έχουμε όλους τους ε, γεωργούς υπόψη στην Επιτροπή. Θέλουμε καλύτερες τιμές και έσοδα για όλους τους γεωργούς ανεξαρτήτως ε, υπηκότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να έχουμε βιώσιμη οικογενειακή γεωργία. Ευχαριστώ. Κύριε Μποβέ, έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε. Σας άκουσα με προσοχή, αλλά δυστυχώς τα λόγια σας ε, δεν ε, βρήκα κανένα σημαντικό σχέδιο. Μίλησατε για αναδιάρθρωση, ενδεχομένως και για απλούστευση. Αλλά ποιο είναι το σχέδιό σας, ένα μακρόπρονο σχέδιο για την επόμενη πενταετία. Εντάξει η απλούστευση, αλλά το θέμα είναι πού πηγαίνει η γεωργία μας, προς τα πού κατευθύνεται. Γιατί όλοι μιλούμε για την κρίση. Όλοι λένε ότι η επόμενη κρίση για το γάλα θα είναι χειρότερη από το 2009 και ταυτόχρονα ποια είναι η λύση που δίνεται, κατάργηση των γαλακτοκομικών προστόσεων. Θα πρέπει να αναλάβετε τι ευθύνε αυτή τη κρίση στο γάλα. Ταυτόχρονα μα λέτε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τι εξαγωγέ. Το άκουσα. Δηλαδή θα αυξήσουμε και τι εισαγωγέ. Τι θα γίνει ότι θα έχουμε 300.000 τόνου κρέατο που θα μα κατακλείσουν από την Βόρεια Αμερική. 1,2 εκατομμύρια κεφάλαια θα οδηγήσουμε στην ε, χρεοκοπία του δικούς μας κτηνοτρόφους, ενώ το 2015 θα έχουμε τη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα στο Παρίσι. Ούτε ε, στο ερώτημα ε, του κυρίου Ντές και του κυρίου Ντεκάστρο μπορείτε να ανταποκριθείτε, γιατί τα δικά του συμφέροντα είναι ενάντια στα συμφέροντα της υφηλίου του πλανήτη μας και του κλίματός μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούιτερμαχτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Πολλά ακούσαμε για το πρασίνισμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει αν θα εξετάσετε ισοδύναμα μέτρα που πρότειναν τα κράτη-μέλη. Πριν από μερικές εβδομάδες ανακαλύψαμε ότι σε τρία διαφορετικά κράτη-μέλη διαπιστώθηκαν κρούσματα γρήπης των πουλερικών. Δεν, δεν φαίνεται σοβαρή έκταση του προβλήματος, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω. Οι κάτω χώρες επέβαλαν κάποια πολύ αυστηρά μέτρα και μάλιστα το Βέλγιο απαγόρευσε τις εισαγωγές, κάτι που είναι απαράδεκτο σε μια ελεύθερη αγορά. Τι σκοπεύετε ε, να κάνετε προκειμένου να διορθώσετε αυτή τη στρέβλωση αγοράς που δημιουργήθηκε από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, όταν μιλάμε για το γάλα είναι σαφές ότι το πρόβλημα είναι συγκυριακό και δύσκολο. Όμως έχουμε και διαρθρωτικό πρόβλημα ή θα έχουμε άμεσα γιατί πριν από λίγο καιρό είχατε πει ότι σε ορεινές περιοχές, δύσκολες περιοχές, μειονεκτικές, θα δημιουργήσει προβλήματα η κατάργηση των ποσοστώσεων. Και εμείς είχαμε κάνει μια έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα. Και είχαμε προτείνει κάποια πράγματα. Η Κομισιόν δεν ανέλαβε δράσεις. Σε μειονεκτικές περιοχές όπως ορεινές θα υπάρξει πρόβλημα μετά την λήξη των ποσοστώσεων. Μέχρι τον Απρίλιο υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι ή ε, δεν θα λάβουμε κανένα μέτρο για το γάλα στις ορεινές περιοχές. Κύριε Σέρντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα για τα προκυπευτικά, για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία. Παρακαλώ να επανεξετάσετε το πρόβλημα, διότι έχουμε και άλλα προϊόντα όπως είναι το γιαούρτι, το κεφίρ, το ξινόγαλα, τη σοκολάτα που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά τα προγράμματα για τα σχολεία ή και οι σούπες. Λοιπόν σκεφτείτε αυτή την πτύχη σας παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το ρωσικό εμπάργο σίγουρα επηρέασε το γαλακτοκοπικό τομέα, αλλά και τα απορροκυπευτικά. Τα μέτρα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου. Οπότε ανακύπτει το πολιτικό ερώτημα πώς θα λύσουμε από εκεί και πέρα το πολιτικό πρόβλημα, γιατί δεν φαίνεται ότι θα σταματήσει το πρόβλημα τέλη Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η ρωσική απαγόρευση, θα παρατείνετε τα μέτρα που όπως είπα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ύψη προτεραιότητα στην ενίσχυση των νέων αγροτών και στην προσέλκυσή του στη γεωργία. Αν δεν λύσουμε όμως το πρόβλημα της τροφικής αλυσίδας, τα προβλήματα δεν σταματήσουν. Το Σώμα των Επιτρόπων ασχολείται με το θέμα αυτό, γιατί έχουμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Με 48 λεπτά το ευρώ αμείβουμε ένα λίτρο γάλακτος Χθε στην Κόρδοβα είδα ένα σούπερ μάρκετ ε, ένα λίτρο γάλακτο σας στοιχεί 48 λεπτά. Πώς να υπάρχει ανταγωνιστικότητα με τις τιμές. Ευχαριστώ κύριος Φλάμαγκεν. Ήρθατε και τα συγχαρητήρια για το νέο σας αξίωμα. Εκφράστηκαν εδώ σε ανησυχίες σε σχέση με την εφαρμογή του πρασινίσματος, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία με το παλιό σύστημα πληρωμών. Κάποιοι θα πάρουν 300 ευρώ ένα εκτάριο, άλλοι 30 για το πρασίνισμα. Ο κίνδυνος είναι ότι στην πορεία θα πει κανείς άμα γίνεται με 30 ευρώ για έναν αγρότη γιατί να μην γίνει και με τον άλλον. Οπότε η Ιρλανδία μπορεί να χάσει κάποια χρήματα αν επιμείνεται σε αυτή τη λύση. Για το γαλακτοκομικό τομέα προφανώς η παρέμβαση είναι απαραίτητη πρέπει να εξεταστεί. Μακροπρόθεσμα υπάρχουν συνεχιζόμενα υψηλά κόστη ζωοτροφών, ενέργειας, ε, οπότε πώς θα βοηθηθούν ε, αναερόβια χώνευση ή όταν έχουμε ε, τομεί που μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων και μακροπρόθεσμα να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα. Μπορεί να γίνει κάτι ε, που θα εξασφαλίζει ε, μόνιμες λύσεις, ε, ενώ άλλες είναι λιγότερο προβλέψιμες. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Καλνιέτε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Φαντάζομαι θα ξέρετε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα 400 εκατομμύρια το δημοσιονομικό πλεόνασμα ε, και ασκήσαμε πίεση να παραμείνει αυτό το αποθεματικό στον προπολογισμό της ε, ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ενώ έχουμε και τα 23 εκατομμύρια που αποφάσισαν για τον γαλακτοκομικό τομέα. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό θα εξασφαλιστεί η επιβίωση για λίγου μόνο, μήνε, μόνο μήνες. Το θέμα είναι πώς θα επιβιώσουμε μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, μετά την 1η Απριλίου. Μπορούμε να ελπίζουμε σε μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το πρώτο εξάμεινο του 2015. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ. Ως Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω από εξ των αγροτών της Λιθουανίας και της Βαλτικής γενικότερα για την, τις γρήγορες αποφάσεις που περιόρισαν κάποιες ζημίες μετά από το ρωσικό εμπάργκο. Επρόκειτο μάλλον για πολιτική απόφαση. Δηλαδή οι περισσότερες επληγήσεις χώρες δεν εγκαταλήφθησαν ήταν ένα μέτρο αλληλεγγύης που έδωσε ελπίδα στον κόσμο στην περιοχή. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Μιλήσατε ότι θα, είπατε ότι θα διατεθούν 200 εκατομμύρια για το άνοιγμα νέων αγορών. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Αλλιώς οι αγρότες μας του χρόνου, γιατί μάλλον και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούν βοήθεια οι αγρότες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις, στην Πολωνία έχουμε στις αποθήκες 700.000 ε, 700 τόνους ε, μήλων. Ένα τμήμα θα πάει στις ασυστητικές αγορές, αλλά 500, 500 με 600 τόνους παραδοσιακά, 500 600.000 τόνους παραδοσιακά στέλναμε προς τη Ρωσία. Αυτά τα μήλα δεν μπορούμε να τα διοχετεύσουμε εξαιτία του εμπάργου. Θα παραμείνουν στις αποθήκες μας, θα σαπίσουν τα μήλα εκεί. Τώρα, ε, έχουμε 10 χώρες που το 2002 διαπραγματεύτηκαν τις ποσοστώσεις και είχαμε αποφασίσει τέλος των ποσοστώσεων το 2007. Το 2003, ήδη χωρίς εμάς, οι 15 χώρες μας απέκλεισαν και μας έδωσαν προτετελεσμένο γεγονότων. Ε, φυσικά, ε, ε οι Πολωνοί Γεωργοί ξεπέρασαν ε, τις γαλακτοκομικές τους ποσοστώσεις, ε, πληρώντας αδρά πρόστιμα απελπιστώντας όμως ότι θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν ε, το πρόβλημα από το εμπάργο. Αλλά δυστυχώς ε, χωρίς την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλοί θα χρειαστεί να χρεοκοπήσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλλερ. Yes. Κυρία Μίλλερ, συγγνώμη. Haben... Κύριε Επίτροπε, είσαστε, χρηματίσατε Υπουργό Περιβάλλοντο και εγώ θέλω να μιλήσω για άλλο θέμα. Αύριο θα έχουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ μια ακρόαση για την οδηγία ΑΝΕΚ μπορείτε να ασκήσετε επιρροή ώστε να ε, ισχύουν τα ίδια μέτρα υπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα σημαίνει για τη Γερμανία ότι από το 2003 οι μειώσεις εκπομπών ε, μεθανίου θα πρέπει να είναι πολύ, ε, οι, μειώσεις θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και οι, οι γεωργοί δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και θα βρεθούν ενώπιον ανεπιλήτων προβλημάτων. Τώρα, η, πολιτική των δασών. Η δασοκομεία είναι πολύ σημαντική παράλληλα με τη γεωργία. Πώς θα κατα... Και τώρα καταρτίζουμε ένα πρόγραμμα. Θέλω να ξέρω θα ελειφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εμείς... Ε, δεν ε, θέλουμε αξιοποίηση ε, ε, καταράκτη όπως λέμε. Ευχαριστώ κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αποδείξατε ότι είστε επίτροπος που τηρεί τις υποσχέσεις του, έτσι φάνηκε με την υπόσχεσή σας και την εφαρμογή των κινήτρων για τους νέους αγρότες. Εγώ κατάγομαι από την Κροατία. Σας, καλώ και σας προσκαλώ στην Κροατία γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσετε λίγο τον, Γεωργό, τον Υπουργό Γεωργίας της Κροατίας που φαίνεται δεν ασχολείται και πολύ με τη Γεωργία. Θα πρέπει να τον παροτρύνετε να ε, λάβει υπόψη ε, τα συμφέροντα των γεωργών. Για παράδειγμα, μέλησε και δεν ζήτησε υποστήριξη για τους παραγωγούς ε, μανταρινών ε, και ροδάκινων από την Κροατία που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργο. Ε, δυστυχώς φέτος χάσαμε 50 εκατομμύρια ευρώ από την αμέλεια του Υπουργού μας, του χρόνου θα χάσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους μηχανισμούς ελέγχων των κρατών μελών για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει τη σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερόν, ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, Λοιπόν, ε, θα πρέπει πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να αναγνωρίσει την ανεπάρκεια της, κοινή της κοινής αγροτικής πολιτικής του 2014-2020 με το πλαίσιο στρατηγικό, το διεθνές και το οικονομικό. Πρέπει να το καταγγείλω. Υπήρξε αντικείμενο μακρών διαπραγματεύσεων να πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί κοινή αγροτική πολιτική όπου κανένα δεν θα ήθελε να εφαρμόσει. Οι μεγάλε δυνάμει αυξάνουν την παραγωγή προσπαθώντας να προστατεύσουν καλύτερα τους γεωργούς τους, όπως έκαναν οι ΙΠΑ με το νέο Farm Bill. Η ΚΑΠ μειώνει τις ενισχύσεις, ενισχύει τους περιορισμούς και δεν επιτρέπει την προστασία των ε, γεωργών κατά τις μειώσεις ε, των τιμών. Ο γαλακτοκομικός τομέας από μόνος του δείχνει τους κινδύνους που διατρέχουμε. Το εμπάρκο του ρωσικού μείωσε επίσης τις τιμές σε ανησυχητικό επίπεδο. Ε, ξέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν την κρίση, θα πρέπει ε, να βλέπουν ότι χάνονται πάρα πολύ με πολλά κέρδη. Λοιπόν, γιατί εφαρμόζεται μια πολιτική που δεν μπορεί παρά να οδηγεί στην καταστροφή, γιατί να επιμένουμε σε αυτήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε γνωρίζω ότι το γάλα μας τρελαίνει τελικά το πρόβλημα του γάλακτος. Οι γεωργοί στη Ρουμανία μιλάνε για απελπιστικά χαμηλές τιμές του γάλακτος. Πρέπει να πολλούν κάτω από το κόστος παραγωγής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και παρόμοια προβλήματα σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μπροστά μας πριν απαλλαχθούμε από τις ε, ποσοστώσεις, ε, τι θα κάνετε, έχετε κάποιο σχέδιο, ούτω ώστε οι γεωργοί που παράγουν γάλα να παράγουν κτηνοτροφικά προϊόντα. Διαφορετικά θα έχουμε ένα τσουνάμι γάλακτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σεμπαστιά ή μάλλον η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε, για την παρουσίαση που κάνατε. Χιλιάδες ζώα ε, βρίσκονται σε χώρους για εντατική αναπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζουν σε φρικτές συνθήκες. Και δεν είπατε τίποτα για την ευημερία των ζώων ήταν παλιά ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή Γεωργίας και για τον Επίτροπο των Ορμόδιων για τη Γεωργία. Και φαντάζομαι για σας τι σχέδια έχετε γι' αυτό. Είπατε ότι θέλετε να προστεύσετε την νομοθεσία. Αυτή είναι η άλλη ερώτηση. Για λιγότερη γραφειοκρατία. Αλλά για κάποια ζώα δεν υπάρχουν κανονισμοί. Δεν υπάρχει νομοθεσία που διέπει την αναπαραγωγή και την εκτροφή των κουνελιών. Θα νομοθετήσετε πάνω σε αυτό ή για άλλα παρεμφερή ζητήματα. Και κάτι ξεχωριστό. Προϊόντα που είναι το φουάγκρα, που οι χήνες εκτρέφονται προς πάχυνση και για την χρήση του σηκωτιού τους. Ε, αυτό είναι ένα επίκαιρο θέμα, κυρίως εποχή Χριστουγέννων. Τι θα κάνετε για να καλύψετε νομικά το θέμα και ιδεοδός να απαγορευτεί η παραγωγή ε, του φουαγκρά. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Σλάιερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κάτω χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη γρήπη των πουλερικών, η οποία μας κοστίζει εκατομμύρια ευρώ και πολλές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πλήγμα που τους χτύπησε τις τελευταίες εβδομάδες με τα κρούσματα της γρήπης των πουλερικών. Σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα. Η γρήπη των πουλερικών όπως και κάποιες άλλες μας ε, μαστίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα προστατεύσουμε τους ε, καταναλωτές, τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα και τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει δυνατότητα θέσπισης ε, ενός μηχανισμού που να εξασφαλίσει την επιβίωση της κτηνοτροφίας παρά τέτοιες επιζωοτίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Νόιτσελε. Κύριε Επίτροπε, πήρατε μία επιστολή υπογεγραμμένη από τέσσερα άτομα με στόχο το πρασίνισμα πριν αρχίσει να το καταστρέψουν. Του... Τις επόμενες μέρες θα πάρετε επιστολές και από άλλους βουλευτές που θεωρούν ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να υφίσταται για τους γεωργούς και στο μέλλον. Και αυτό θα γίνει μόνο αν έχει καλή νομιμοποίηση ο πρώτος πυλώνας. Και το πρασίνισμα είναι πολύ σημαντικό εδώ. Μία ερώτηση λοιπόν ε, θέλω να σας κάνω για άλλο θέμα όμως. Ξέρετε το ε, έγγραφο της επιστημονικής υπηρεσίας της Γερμανικής Βουλής που λέει ότι ε, αν ε, εγκριθεί ε, το TTIP θα έχουμε πρόβλημα ε, με προϊόντα ε, και που χρησιμοποιούν μεταλλαγμένα. Πώς θα γίνει η σήμανση. Θα έχουμε προβλήματα ως προς αυτό με την συμφωνία TTIP. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Ευχαριστώ λέει κυρία Ριμπέρα. Έχουμε πρόβλημα με το γάλα και τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Ξέρουμε ότι καταβαραθρώθηκαν οι τιμές γάλακτος και οι προοπτικές είναι μάλλον ζωφέρες. Οπότε μάλλον θα επαναληφθεί η κρίση του 2009. Μάλιστα, το ρωσικό εμπάργο μας έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει το πλεόνασμα της παραγωγής και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο γάλα ήταν απολύτως αποτελεσματικά. Κύριε Επίτροπε, είστε έτοιμος για διαπραγμάτευση και για θέσπιση κάποιων μέτρων ρύθμισης αγοράς γάλακτος, όπως πρότεινε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ο κύριος Νταντά. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω και στις Αζόρες, σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή της Πορτογαλίας, για να δείτε και η πόσο σημαντική είναι η γεωργία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, για τη χωροταξία, αλλά για την καταπολέμηση των προβλημάτων που δημιούργησε το ΠΟΖΕΙ, το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Είστε έτοιμος να αναθεωρήσετε το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας ε, και για την προθυμία σας για συζήτηση. Και εγώ έχω ένα σχόλιο για το γάλα που αναφέρθηκε από πολλούς προλαλήσεντες. κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για την Ευρώπη. Η ερώτησή μου αφορά την διακοπή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Δυστυχώς αυτή η διακοπή ευνοεί ορισμένους και πλήττει άλλους. Πώς θα αξιολογήσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα κάποιων αποφάσεων και μερικές φορές ε, ε, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ε, η διακοπή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων σκόπο, σκοπό είχε την βελτίωση της αγοράς γάλακτος, όχι την εξώθηση στη χρεοκοπία των κτηνοτρόφων. Η γαλακτοπαραγωγή για μερικές περιοχές και για μερικούς παραγωγούς είναι η μοναδική ε, λύση επιβίωσης. Δεν υπάρχουν άλλες βιώσιμες εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Νταντσίλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με την ε, υπερβολική αστάθεια των τιμών στο γαλακτοκομικό τομέα δεν πλουτίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί, αλλά οι μεταποιητές του γάλακτος. Και με την ε, κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2015, θα πρέπει να βρούμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων των παραγωγών και των συμφερόντων των μεταποιητών ή των ε, σούπερ μάρκετ, των λιανεμπόρων που αποφελούνται σε τελική ανάλυση από αυτή την κατάργηση και την αστάθεια των τιμών. Τι μέτρα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθώσει την ανισορροπία. Πρόεδρε, ε, ε, τελικά είναι δοκιμή αντυχής και πνευματικής αντυχής για τον Επίτροπο. Αρχίζω να τον λυπάμαι. Λοιπόν, βλέπετε 30 τέτοιε παρεμβάσει των λεπτού πρέπει να επαναξεταστεί. Δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθο, ούτε μπορούμε να εκφραστούμε ειλικρινά. Επ' αυτή τη βάση να πω επίτροπε ότι καλωσορίζω προσπάθειες σα για απλούστευση. Θα σα στείλω μια έκθεση που ετοίμασε η κοτική κυβέρνηση και είχα στείλει στον προκάτοχό σα που αφορούσε την ε, μείωση της γραφειοκρατίας. Και μπορούμε να σας στείλουμε και στους υπόλοιπους ε, να δείτε τι προσπάθειες πρέπει να κάνει ο Επίτροπος ώστε τελικά τα λόγια του να γίνουν έργα όσον αφορά την ε, απλούστευση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Πρέπει να πω ότι υποσχέθηκατε προλίγου ότι δεν θα φύγετε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Είπατε ότι δεν θα αφήσετε μάλλον τους παραγωγούς στη μοίρα τους. Έχω ερωτήσεις. Τι θα κάνετε για να σταματήσει ε, η διακύμανση των τιμών στον τομέα το γαλακτοκομικό μετά την κατάργηση των ε, ποσοστώσεων. Ίσως αν θέτουμε συνεχώς το ερώτημα αυτό θα πάρουμε τελικά απάντηση. Επόμενο ερώτημα. Οι γεωργοί δεν είναι σε θέση να πωλήσουν τα προϊόντα τους ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για να αποζημιωθούν γι' αυτό. Τι προτεραιότητα θα δώσετε όσον αφορά την τοπική παραγωγή των τοπικών εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δες που είναι και ο τελευταίος στον κατάλογο των ομιλητών. Είπατε κάτι συγκεκριμένο ότι τα επόμενα δύο χρόνια στο πρασίνισμα δεν θα υπάρχουν κυρώσεις. Αυτή η δήλωση ε, βρίσκει σύμφωνο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάλιστα. 40 βουλευτές συνολικά έλαβαν το λόγο στην ανταλλαγή αυτή απόψεων με τον ε, Επίτροπο. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί ήσασταν υποδειγματικοί όλοι στην τήρηση της, ε, του χρόνου ε, και λυπούμε που σας ε, έβαλα σε τέτοιο κλειό και λυπούμε και για την ταλαιπωρία του Επιτρόπου αλλά αυτά έχει η θέση σας. Τέθησαν πολλές ερωτήσεις, πολλές έμοιαζαν αλλά θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ όσον αφορά το βόηο κρέας καταρχάς να πω ότι είναι τεράστιο το ζήτημα όσον αφορά τη μεταβολή των τιμών του βοηού από Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο του 2014 συγκρίση με την παρόμοια περίοδο του 2013 αν γέννη είχαμε αύξηση των εξαγωγών 23,2%. Ε, θεωρώ ότι μπορούμε να, πηγαίνουμε, να πάμε πολύ καλύτερα, να βρούμε και άλλες αγορές και να διαθέσουμε πόρους σημαντικούς για την πρόθεση των γεωρικών προϊόντων γνωρίζουμε ότι στις διάφορες εμπορικέ διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούμε στα πλαίσια του TTIP είναι σημαντικό τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και που είναι σημαντικές οι προδιαγραφές που τονίσατε να υποστηριχθούν. Το γνωρίζω, το είπα και αρχικά. Δεν θα θυσιάσουμε την ποιότητα και θα προσέξουμε τα ευαίσθητα προϊόντα, κυρίω το βόλιο κρέα, όσον αφορά το μερίδιο τη αγορά και να παραμείνουν οι τιμέ που είναι καλέ για του γεωργού, όσον αφορά το γάλα. γίνονται σοβαρές οι αλλαγές στον τομέα λόγω των θεσπιστέντων κανόνων και της πολιτικής. Το 2008 που είπαμε θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις γαλακτοκομικές το 2015 λόγω κλιματολογικών συνθήκων σε κάποιες χώρες είχαμε αύξηση του 5% όσον αφορά τον όγκο της παραγωγής του γάλακτος. Βέβαια αυτό θα έχει αντίκτυπο, είναι σίγουρο. Ακόμα και κάποιος που έχει ελάχιστες γνώσεις ε, οικονομικών ε, το γνωρίζει ότι θα είναι ευμετάβλητες οι τιμές του γάλακτος. Να καταλάβουμε ότι η μέση τιμή ενός λίτρου γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 30 cents. Δεν αντιμετωπίζουμε ακόμα μεγάλη κρίση. Ε, έχουμε ξεφύγει από τις πολύ ψηλέ τιμές και ξέρουμε ότι είναι και πόσο είναι το κόστος παραγωγής ε, είναι κάτι προβληματικό στα κράτη-μέλη. Αλλά έχουμε και μείωση της τιμής του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες και σε επίπεδο κρατών μελών ίσως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εισρωής που ε, προέρχεται από τη μείωση του κόστου ενέργεια και αυτό να μετακυλιστεί στον παραγωγό, αυτή η μείωση του κόστου, και στον κόσμο που χρειάζεται να μειώσουν το κόστος των ζωτροφών, των ε, λοιπασμάτων κλπ. Το κόστος τη εκμετάλλευση εν γέννη. Και αυτό να το έχετε υπόψη μέλη του Κοινοβουλίου και παρακαλώ να μου δώσετε κάποιε πληροφορίε, Διότι θα εξετάσει το θέμα και σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά στην κοινή οργάνωση της αγοράς του γάλακτος έχουμε αρκετά εργαλεία να το αντιμετωπίσουμε το θέμα του γάλακτος. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες, εισακούω τις ανησυχίες σας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία στην αγορά. Εκεί που μπορούμε να παρέμβουμε ταχύτερα, σε ένα πιο πρώιμο στάδιο από ό,τι κατά το παρελθόν. Αλλά σίγουρα ανταποκρινόμεθα όσον αφορά την απαγόρευση τη ρωσική Υπάρχουν χώρες που έχουν υποφέρει περισσότερες από τις άλλες. Στην Πολωνία, πραγματος χάρη, αναφέρθηκε 25% μείωση των εξαγωγών είχαμε, αλλά 7,2% μείωση στις τιμές. Έχουμε αυτά τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη που μας έρχονται κάθε μήνα. Όταν πέντε στοιχεία μείωση της τιμής 20% δεν είναι σωστές. Οι πολωνικές αρχές μας λένε τελευταία μείωση της τιμής ε, του γάλακτος ήταν 7,2%. Στις βαλτικές χώρες είχαμε 22,2% μείωση στην Εστονία 20,3% στη Λετωνία και 12,6% μείωση των εξαγωγών πρόσφατα στις βαλτικές χώρες και παρόμοια μείωση των τιμών. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν ε, όσον αφορά τις χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα με μικρά ποσά για να δείξουμε αλληλεγγύη σε γαλακτοπαραγωγούς και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το θέμα με τη Φιλανδία όπου εκεί ζητήσαμε από τις αρχές της Φιλανδίας να μας δείξουν πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε μία απόφαση να τους υποστηρίξουμε. Είμαστε ακόμα συνομιλίες. Κυρία Ντότς, χτες όσον αφορά την αγορά του γάλακτος η τιμή έπεσε κατά 1,1 σέντ. Δεν ήταν τεράστια η μείωση, αλλά είχαμε κάποιες αυξήσεις στην τιμή του βουτύρου και των τυριών στην ίδια αγορά Άρα θα πρέπει ίσως να εξισορροπήσουν ε, τα διάφορα προϊόντα το ένα το άλλο. Τώρα όσον αφορά το γάλα, γιατί σαν πολλά ερωτήματα. Ε, σίγουρα θα έχουμε βραχυπρόθεσμα πολύ μεγάλη μεταβολή των τιμών, θα παρακολουθούμε και είναι και στην κατάσταση, έχουμε μηχανισμούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά μην τελικά δημιουργήσουμε την κρίση όταν δεν υπάρχει με τα λόγια. Θα αντιμετωπίσουμε τι κρίσει από το εμπάρκο της Ρωσίας στα προεκριστικά και στο γάλα. Ε, και έχουμε εφαρμόσει στο μέτρο του δυνατού τα σχετικά μέτρα για τους συγκεκριμένους τομείς. Όσον αφορά το TTIP, πρώτη ερώτηση ήταν αυτή, αφορούσε τις συνομιλίες TTIP. Είπα επανειλημμένα ότι θα υπερασπιστώ τη Γεωργία στα πλαίσια των λόγων διαπραγματεύσεων. Σαν Επίτροπος ε, για τη Γεωργία θα εμπλακώ στις ε, διαπραγματεύσεις και θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Μάλστρομ ώστε να έχουμε ισορροπημένη συμφωνία το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο δεν είναι κάτι θα διαπραγματευτούμε και κυρίως οι κοινωνικές επιλογές δεν είναι επιτάπητος προς διαπραγμάτευση. Το TTIP δεν θα οδηγήσει σε πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου στη γεωργία και όπως σας είπα θα έχουμε υπόψη μας τα ευαίσθητα προϊόντα. Ξέρω ότι είναι σημαντικό ο Επίτροπο Μάστρομ να μπορεί να, το πει, να τα πει αυτά και να θέσει τι θέσει διαπραγματευτικέ καθαρά και αυτό θα κάνει στο μέλλον, ούτω ώστε ε, να ε, τελικά να μην υπάρχει τόσο μεγάλη μυστικότητα. Λοιπόν, αυτό που είπε η κυρία Γκαρσία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει παραλληλισμός μεταξύ των διαφόρων τομέων που διαπραγματευόμαστε στις συμφωνίες που κάνουμε και η πρόσβαση στις αγορές και οι γεωγραφικές ενδείξεις θα λαμβάνονται υπόψη. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις ήταν αυτή η απάντηση. Λοιπόν, τώρα για τους κοινούς βοσκότοπους στην Ιρλανδία. Λοιπόν, και στα πλαίσια της ανάπτυξης υπαίθρου στην Ιρλανδία, εμείς αναλύουμε τη συγκεκριμένη πρόταση που υπάρχει και είμαστε διαπραγματεύσεις με τις Ιρλανδικές αρχές, διότι μας στείλανε μια επιστολή και δώσαμε σχετική απάντηση με αυτό. Το σχέδιο πρόγραμμα αναπτύξης υπαίθρου προβλέπει ότι για να υπάρξει πρόσβαση στο πρόγραμμα θα πρέπει οι γεωργοί να έχουν προβάλει ένα σχέδιο για την χρήση των κοινών βοσκοτόπων και όχι μεμονωμένα, όλοι μαζί με τουλάχιστον ε, εκείνοι που έχουν 50% του κοινού βοσκοτόπου και θα πρέπει τελικά να προστατευτούν και οι λόφοι ε, που χρησιμοποιούνται ε, διότι συμβάλλουν στη βιοπικιλότητα. Θέλουμε όμως να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η γη και σε μελλοντικό σχήμα γεώργο παραγωγικό και να βρούμε μια λύση ούτως ώστε οι μεγαλύτεροι κοινοί βοσκότοποι και οι γεωργοί που χρησιμοποιούν του βοσκότοπου να ζητήσουν υποστήριξη για το περιβάλλον και να υπάρχει συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών αυτών βοσκοτόπων. Τώρα, για τη ρωσική απαγόρευση για τα απορροκυπευτικά. Ο Πολωνός Ευρωβουλευτής το έθεσε αυτό στο πρώτο πακέτο, 87% των αιτήσεων ήρθαν από την Πολωνία για τα προκυπηστικά. Μόνο 18% του ποσού που κοινοποιήθηκε τελικά απορροφήθηκε για τα μέτρα που εφαρμόστηκαν. Δεν ξέρω τι συνέβη μεταξύ της ημερομηνία των αιτήσεων και μέχρι της απορρόφησης των ενισχύσεων. Πολλοί γεωργοί απουσίαζαν στη συγκεκριμένη περίσταση. Και είχαμε ένα δεύτερο πακέτο που κάποιοι γεωργοί ήθελαν ξανά να υποβάλουν αίτηση. Αλλά η πολωνική αντιπροσωπεία στο δεύτερο πακέτο. Ε, μάλλον έχουμε 18.750 τόνους για μήλα και ε, ε, αχλάδια. Και αποσύρθηκαν πάρα πολύ, 90% πήγανε για ζωοτροφές 90% από αυτά, από το πλεόνασμα. Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα μήλα σε κάποια κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένη τη Πολωνία. Και εξακολουθούμε να εξετάζουμε, να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Και αυτό ισχύει συγκεκριμένα ειδικά για την ε, Πολωνία. Μετά, για την γρήπη των πουλερικών, υιοθέτησε τρει αποφάσεις κατεπίγουσας ανάγκη για τη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθορίζονται οι περιοχές όπου είναι που περιορισμού στην κτηνιατρικού εφαρμόζονται οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχουν στόχο το ώστε να ελεγχθεί η ζωονόσος και να μην διαδοθεί, διότι είναι πολύ μεταδοτική αυτή η ασθένεια. Για να ελέγξουμε λοιπόν τη διάδοση του ιού, στα τρία κάτι μέλη εφαρμόσαμε τα μέτρα προβλέπονται από το Συμβούλιο. Τα μέτρα συμπεριλαμβάνε το να σκοτωθούν τα πουλερικά, να πρέπει να υπάρχουν ζώνη που ελέγχονται και θα πρέπει να εφαρμοστούν υγειονομικά μέτρα και επίση ενημερώσαμε και τα άλλα κράτη-μέλη σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη-μέλη μη Ευρωπαϊκή Ενώση και διεθνεί οργανισμού για την όλη κατάσταση όσον αφορά την ασθενεία και ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα τελικά λειτουργούν, φέρνουν αποτελέσματα, αλλά σίγουρα αυτό θα το εξετάζω και θα σα ενημερώσω σχετικά και θα ενημερωθώ όταν θα πάω στην Ολλανδία την Πέμπτη. Ξέρω ότι έχει πληγεί όλο ιδιαίτερο η Ολλανδία από την ε, γρήπη των πουλερικών όσον αφορά τι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει στι Αζόρε και κατάργηση εν γέννη των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Αυτό είναι κάτι που ε, αναφέρεται πολύ συχνά στις συζητήσεις, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες ε, το μέσο της οδού. Το 2008 υιοθετήθηκαν οι κανόνες. Ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη συμμορφώθηκαν με τους κανόνες αλλά έχουμε μια δύσκολη κατάσταση κάποια κράτη-μέλη σε αυτή τη φάση, διότι σχεδιάζουν εκ των προτέρων για την κατάργηση των ποσοστώσεων και ίσως να το κάνουν πολύ πρωιμά αγοράζοντας παραπάνω γελάδες, να βάζουν περισσότερα στοιχεία για την παραγωγή γάλακτος. Σε κάποια κράτη-μέλη, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, ε, υπάρχουν πολύ ευμενείς κλιματολογικές συνθήκες, οπότε μπορούν να ε, παράγουν το γάλα σε πολύ καλές τιμές και να το πολλούν και οι γεωργοί ε, αποφάσισαν να συνεχίσουν την παραγωγή και τους ζητάω. Μέσω ημών στους κοινοτρόφους σας λέω να λάβουν τα αναγκαία μέτρα τώρα ώστε να καταλάβουν ότι δεν θα υπάρχει αλλάξη στο, θα, αλλάξει το καθεστώς ε, όσον αφορά τις ποσοστώσεις. 31 Μαρτίου θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις και θα πρέπει άμεσα να γίνει δράση, να λέω του δράση και τα κράτη-μέλη και οι γεωργοί. Τώρα, υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπο που είχε αυτό στις ε, Αζόρες. Θα εξετάσω λοιπόν το όλο πρόγραμμα για τις Αζόρες να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα που αναφέρατε συγκεκριμένα με αυτή την περιοχή ε, και τις ιδιαίτερες περιστάσεις που μου παρουσιάσατε. Η κατάσταση λοιπόν ε, για τις ποσοστώσεις θα είναι αυτή που περιέγραψα. Και ίσως θα μπορούσα να σας βοηθήσω για την άψη της υπαίθρου, να βοηθήσουμε τους ε, γεωργούς μέσω της αναδιάθρωσης ε, ήταν αύξηση πέφτου αζόρεστο. το σύστημα για το σχολικό γάλα ήταν αντικείμενο εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εργασίας δεν ολοκληρώθηκε ακόμα ε, για το 2015. 16 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί και εκεί θα έχω τις προτεραιότητες και θα τις θέσω σώμα των επιτρόπων και θα δούμε κατά πόσο θα συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα του σχολικού γάλακτος δεν πιστεύω ότι θα συμπεριληφθούν οι ελιές εάν ε, γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε πολύ λίγα χρήματα και έχουμε και το αποθεματικό από την κρίση και ήθελα να το προστατεύσω αυτό και το ανέφερα προηγουμένω. Και η τροποποιητική η διορθωτική επιστολή της 15 ε, Οκτωβρίου του 2015 ε, Οκτωβρίου του προπολογισμό δεν θέλει να ε, ε, θέλει να βοηθήσει να αντιμετωπίσουν διακύμαση των τιμών και αυτό θα έχω το μέσο στη διάθεσή μου το 2015 και συνεργάζομαι πολύ στενά με την Επίτροπο τη Γεωργίευα, την υπεύθυνη για τον προπολογισμό να συνεχίσουμε να έχουμε τα 433 εκατομμύρια ευρώ για το 2015 αυτό που είπατε, λόγω της διακύμασης των τιμών, λόγω, λόγω της κατάργησης των ποσοστώσεων και λόγω γεωργικών προβλημάτων και όχι πολιτικών. Τα ανέφερα στις ακροάσεις ότι θα κάνω κάτι από αυτού, και έχω σημειώσει σημαντική πρόοδο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του προπολογισμού και είμαι σίγουρο ότι εκείνοι που εμπλέκονται στι διαπραγματεύσει του προπολογισμού, σα οι νομοθέτε, θα είναι φίλοι μου όσον αφορά τα διαμόρφωση συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Άλλα θέματα. Ε, όσον αφορά το πρόγραμμα για την άψη πέθρου, ενημέρωση. Λόγω του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου και των σχετικών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο και ο κανονισμό δεν υπεγράφει παρά μόνο τον Ιούλιο, υπάρχει μια καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή του προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου. Όπω προανέφερα στην ομιλία μου, δεν θα επηρεάσει κάθε κράτο μέλο στον ίδιο βαθμό. Θα εξακολουθήσουμε τι προσπάθειέ μα και από τώρα μέχρι 1η Ιανουαρίου και Μάιο όλα τα προγράμματα θα εγκριθούν. Όσον αφορά το κάτω μέσο που γνωρίζετε καλύτερα, νομίζω ότι υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο που θα συμφωνηθεί, αλλά υπάρχει και περιφερειακή διάσταση και έχετε πολλούς ε, τομεί προγραμματισμού, περιοχέ προγραμματισμού σε μια χώρα όπω η Γαλλία που θα έχουν διαφορετική εφαρμογή ανάλογα με την περιοχή και την περιφέρεια. Και το εθνικό πλαίσιο αφού δημοσιευθεί, θα δημοσιευθεί μέχρι τέλο του έτου, ελπίζω και στην περίπτωση τη Γαλλία τότε θα μπορούμε να ε, δούμε τις αντιδράσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπου έχουμε ένα μεγάλο κάτω μέλος έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Όταν έχουμε μόνο ένα πρόγραμμα αναπτύξεως υπαίθρου όπως τα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει συνεχής δουλειά που γίνεται. Και ελπίζουμε τελικά ότι μέχρι τέλος Μαΐου του 2015 ότι όλα θα έχουν δρομολογηθεί σωστά η αλλαγή του κλίματος και η στατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Προσβλέπω στην υποστήριξη του εισηγητού ε, όσον αφορά τα δασοκομεία. Συνεχίζεται η δουλειά και ελπίζω να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα αποτελέσματα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το πώς έχουμε προχωρήσει. Έχουμε ένα σχέδιο στρατηγικής για τη δασοκομεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά θέλω να ακούσω τις απόψεις της συγκεκριμένης Επιτροπής ε, πριν ε, έχουμε τελική στρατηγική και βέβαια η αλλαγή του κλίματος ε, Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αναγνωρίθηκε στο πακέτο της ενέργειας και το κλίμα η σημασία που έχει να έχουμε απορρόφηση του άνθρακα μέσω της δασοκομείας και αυτή η απόφαση έχει αποσαφινιστεί λόγω του προγράμματος εργασίας που απαιτείται και λόγω της συνεισφοράς που θέλουμε να έχει η Γεωργία, ούτως ώστε να προσαρμοστούν οι εκπομπές, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε ταυτόχρονα ότι εξισορροπείται με την αναγκαία ασφάλεια των τροφίμων, που είναι κάτι που ανέφερα εξ Ξέρω ότι δεν έχω καλύψει τα πάντα, αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε να διστάσω στον φίλο μου, τον κύριο Μακάρτη, όσον αφορά του ε, ελέγχου και τι επιθεωρήσεις. Και απαντάω και στον κύριο Ντά. η έλεγχη είναι κάτι που είναι τεράστιο πρόβλημα για εκείνου που είναι δικαιούχοι, οι ετούντε. Και εκεί έρχεται και η απλούστευση για το 2015. Λοιπόν, σα εθαρρύνω να μα δώσετε προτάσει, αλλά και εμπειρίες ε, των δικαιούχων. Το λέω σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου αυτό και με τα χαρά να εξετάσουμε προσεκτικά όλα αυτά και να λάβουμε υπόψη όσο δυνατόν περισσότερε, αυτέ που είναι λογικέ βέβαια και μπορούν να βελτιώσουν το εφιστάμενο σύστημα. Τέλο, Πρόεδρε, διότι ξέρω ότι θέλετε να λήξει η συνεδρία. Όσον αφορά τις κυρώσει για το πρασίνισμα, το ελεγκτικό συνέδριο ξέρει ποια είναι η θέση. Η πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά το πρασίνισμα, αλλά και αν η πολιτική δεν εφαρμοστεί ορθά, Βεβαίω θα υπάρξει μείωση των πληρωμών προ το δικαιούχο, αλλά σε περίπτωση όπου υπάρχει κάποιο σφάλμα που έχει διαπράξει ο δικαιούχο όσον αφορά ε, του ποινικούς ε, χώρους ε, δεν θα υπάρχει για την επόμενη διετία ακύρωση που θα εφαρμόζεται. Και το γνωρίζει αυτό πολύ καλά το ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστούμε. Φυσικά ήταν αδύνατο να δώσετε αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Πάντως κύριε Επίτροπε, ε, περιμένουμε να αναλάβετε πολύ δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις για το πρασίνισμα, το γάλα, το εμπάργκο, το TTIP. Πάντως ε, έχετε δώσει την εντύπωση ότι είστε πολύ δυνατή προσωπικότητα, έντονη προσωπικότητα. Ξέρετε τώρα ποιες είναι οι προσδοκίες μας, τι περιμένουμε από εσά και ελπίζουμε να δράσετε αναλόγως. Σας εύχομαι και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος που θα είναι δύσκολος χρόνος. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή και στο μέλλον. Χαιρετίζω και τον εκπρόσωπο της ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ. Θερμά ευχαριστώ και πάλι κύριε Επίτροπε για τη διαθεσιμότητά σας. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία για μια δύσκολη εποχή και για έναν περίπλοκο τομέα όπως είναι η γεωργία για την επόμενη πενταετία. Ε, σας μοιράσαμε ένα σημείωμα με τις αποφάσεις των συντονιστών. Ελπίζω να λάβατε γνώση. Η αυριανή συνεδρία, όπως σας είπα, ακυρώθηκε. Δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Και ελπίζω, κύριε Επίτροπε, στην επόμενη μας συνάντηση να έχουμε περισσότερο χρόνο για συζήτηση. Θα ήθελα τώρα να σας προσκαλέσω όλους ε, σε μία σεμνή τελετή, σε μία δεξίωση ε, εν ώψη και των Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ευχαριστώ και πάλι τους διερμηνείς, να είστε καλά. Πολλές ευχές σε όλους και καλές γιορτές.